Good afternoon, dear colleagues. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Μια και ο πρόεδρος μας έχει μπλοκαριστεί κάπως εκτός κτηρίου, θα ξεκινήσω εγώ τη συνεδρίαση και ελπίζω στο μεταξύ να καταφτάσει και εκείνος. Θα ήθελα να εγκρίνουμε πρώτα την ημερήσια διάταξη και να σας αναγγείλω και κάποιες αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Το σημείο 18, ψηφοφορία ε, της έκθεσης Γκέντς. Ε, θα γίνει αύριο το πρωί από τις 11 παρατέταρτο μέχρι τις 12.30. Μετακινείται δηλαδή λίγο πιο νωρίς. Και η συνεδρία των συντονιστών που θα γίνει και κλεισμένα το θηρό θα αρχίσει 12.30. Έκθεση Βίξτρομ θα ψηφιστεί το απόγευμα, το σήμερα 13 δηλαδή, από τις 4 και 4 μέχρι τις 5 και το σημείο 21 επίσης ε, αναβάλλεται για την επόμενη μας συνεδρίαση. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρώ ε, ως εγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη. Έχω αρκετές ε, ανακοινώσεις. Ε, δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Καταρχήν, διορισμός εισηγητών. Κυρία Γκαμπριέλ, από το ΕΛΚ έχει διοριστεί η συγκήτρια για δύο εκθέσεις για την επανεισδοχή ε, ατόμων που μένουν χωρίς έγκριση και πρόθεσμες ε, ε, θεωρήσεις από το Πράσινο Κρατήριο, κυρία Σόμερ ε, από το ΕΛΚ για το Smart Borders Package, το πακέτο για τα ευφύ για, εισηγητής για τη Europol. Η κυρία Ματιέ είναι εισηγητή στην πρόταση Ευρωπαϊκής, της, του κανονισμού προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ΣΕΠΟΛ. Ο κύριος Έγγελ του ΕΛΚ έχει οριστεί εισηγητή στην πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας 2008-114 για τι κρίσιμε υποδομέ. Και η κυρία Σαρτζεντίνη, ε, συντάκτρια γνωμοδότης προς την Επιτροπή Ήτρε, προς μια ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή στρατηγική για το cloud computing για την Και Ο κύριος Τεγιόγκ θα είναι συντάκτης γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Πολιτισμού για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Επίση να σα επενθυμίσω ότι η ψηφοφορία για το πρόγραμμα δικαιοσύνη για το 2012-2014 θα λάβει η χώρα αύριο στι 9 σε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Σε άλλη αίθουσα όμω στην μεγάλη αίθουσα του τρίτου ρόφου του άλλου κτηρίου. Και υπό επιτροπή Ανθρωπίων Δικαιωμάτων οργανώσει 29 Νοεμβρίου ανταλλαγή απόψεων για την συνοχή εξωτερικών και εσωτερικών απτυχών στην πολιτική θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συμμετοχή του κ. Μόρτεν Κλέρουμ, του Διευθυντού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και φυσικά είστε προσκεκλημένοι σε αυτή την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Λίμπε και Γιούρι. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω θερμά την Επίτροπο Μάλμστρομ, να της εκφράσω την ε, χαρά μας ε, για τη σημερινή αυτή συνάντηση. Θα εξετάσουμε ζητήματα προτεραιότητας στα, στις εσωτερικές υποθέσεις και θα σας δώσω το λόγο προκειμένου να έχουμε αρκετό χρόνο μετά και για τις ερωταπαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξαναέρχομαι στην Επιτροπή σας ε, και που μου δίνετε ευκαιρία να εξετάσουμε κάποια σημεία ε, από το πρόγραμμα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων από τις εργασίες του τομείς αυτούς. Πριν από τρία χρόνια, περίπου την ίδια μέρα, εγκρίναμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Πολλές δράσεις ε, έχουν ήδη υλοποιηθεί, χάρη και στη δική σας άοκνη προσπάθεια και σημαντική συνεργασία και σημειώνουμε πρόοδο σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενό χώρου ασφάλεια, δικαιοσύνη και ελευθερία. Θα ήθελα να σα ε, απαριθμίσω ορισμένα θέματα που ήδη έχουν ε, ολοκληρωθεί ή που θα ολοκληρωθούν ως όνομα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το πακέτο για το άσυλο. Πιστεύω ότι πραγματικά θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ε, την πολιτική συμφωνία για όλα τα νομικά μέσα μέχρι τα τέλη του έτου, αρκεί να κρατήσουμε αυτή την πολιτική όθηση που έχει δημιουργηθεί χρειαζόμαστε μια τέτοια πολιτική συμφωνία πριν το νέο έτος. Πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικός αυτό το στόχος για την υλοποίηση της επιτεύξη της πολιτικής συμφωνίας. Ήταν αμέριστη συνεργασία ε, και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαριστώ τους και οδησηγητές. Καταρχήν έχουμε συμφωνία για τις ε, ε, συνθήκες υποδοχής και μια συμφωνία και για το Δουβλίνο. Σε ό,τι αφορά τις οδηγίες για τα διαδικαστικά έχουμε εκεί και πρόοδο και επίσης την οδηγία για το Eurodac θα το συζητήσετε δεν κάνω λάθος, αυτό το απόγευμα ή αύριο. Βασικός βέβαια στόχος είναι να έχουμε μια, ε, ένα κοινό, ε, μια κοινή πολιτική ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να δίνουμε αρκετή προστασία, επαρκή προστασία σε όσοι τη χρειάζονται. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τα μέχρι τώρα επιτεύγματά μας και θα πρέπει ε, να έχουμε ένα ε, κοινούς κανόνες, ε, κοινέ διατάξεις και κοινά αποτελέσματα. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερη υπερήφανοι για αυτά που έχουμε επιτύχει σε αυτή τη θητεία και θα είναι πραγματικά ιστορικά αυτά τα επιτέγματα γιατί πραγματικά με ευθύνη και αλληλεγγύη μπορούμε να υλοποιήσουμε τους στόχους. Είχαμε επικοδομητικές συμφωνίες μεταξύ των θετισμικών οργάνων. Βέβαια, η Κομισιόν δεν συμφωνεί με, λυπάται για την θέση του Συμβουλίου, αλλά θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε και πού μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβαστικέ προτάσεις, να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε ένα γνήσιο σύστημα ευρωπαϊκό, ώστε να εξασφαλίσουμε εύρυθμη λειτουργία του Σέγγεν, δηλαδή ελεύθερη διακίνηση των προσώπων χωρίς ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα. Κάτι που ε, εκτιμούν ιδιαίτερω οι πολίτε, γιατί είναι αυτό αποτέλεσμα τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τουλάχιστον ε, υπό το πρίσμα των Ευρωπαίων πολιτών. Λυπάμαι που το Συμβούλιο ακόμη δεν κατάφερε να καταλήξει συμφωνία για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και την, προσχώρησή τους, ε, την πλήρη προσχώρησή του στον χώρο του Σέγγεν. Βέβαια, να πω και στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν. Σε εκείνου βρίσκεται το μπαλάκι. Χρειαζόμαστε μία προσέγγιση που θα είναι και νομικός και εμπράκτος εφικτή. Τώρα, για το ΣΥΣ 2 να πω δύο λόγια. Συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν 2. Τα τελευταία χρόνια έχουμε σημαντικές ε, πρόοδους και τελικά παρά τις ταλαιπωρίες επανήλθαμε στο σωστό δρόμο. Είχαμε ε, και ε, την αίσια έκβαση του, δεύτερου, του δεύτερου συστήματος δοκιμής και πιστεύω ότι το σύστημά μας είναι εύρωστο. Παρά την ετοιμότητα όμως σχεδόν όλων των κρατών μελών, κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να αναβάλουμε την ε, θέση σε λειτουργία μέχρι ότου όλα τα κρατημέλη και ιδιαίτερα η Φιλανδία έχουν ε, ετοιμάσει πλήρω τα εθνικά του συστήματα. Πήγαμε στη Φιλανδία με τι υπηρεσίε πριν από δύο εβδομάδε και εκεί ε, καταλήξαμε σε διάφορε προτάσει μετριασμού του κινδύνου και με του Φιλανδού ε, καθορίζουμε το χρονοδιάγραμμα για να δούμε τι αντίκτυπο θα έχουν οι καθυστερήσει. Πάντω θα δώσουμε στα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία πλήρη αξιολόγηση των επιπτώσεων πριν το Συμβούλιο Υπουργών ε, Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων ε, του Νοεμβρίου. Και φυσικά μας ενδιαφέρουν και οι μεταναστευτικέ ροέ στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στη διέλευση από τη θάλασσα, Φέτος είχαμε μικρότερο αριθμό από ό,τι πέρυσι. Παρ' όλα αυτά είχαμε πολύ σημαντικές αφήξεις στη Μάλτα, τη Λαμπεντούζα και αλλού. Και δυστυχώς ε, εξακολουθούμε να έχουμε απώλειες ζώων στη Μεσόγειο με μικρά σκάφη που ναυαγούν. Θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τα κρατημέλη για να σωθούν ζωές και στην Ελλάδα και αλλού. Φυσικά έχουμε την έκθεση του Γιώργου Σόρνου του κυρίου Μούλτερ θα βελτιώσουμε την επιτήρηση ακόμη και στα μικρά σκάφη ώστε να σώσουμε περισσότερε ανθρώπινε ζωέ και ευελπιστούμε ότι θα καταλήξουμε ω ονούπο σε συμφωνία για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τι σχέσει με τι γειτονικέ χώρε, και αυτέ είναι θεμελιώδει και έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά την εταιρική σχέση κινητικότητα με το Μαρόκο. Είχαμε τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων τον Οκτώβριο και με την Τινησία ε, έχουμε συμφωνήσει με τις αρχές για ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων ε, σε, δύο, σε καμιά δύο εβδομάδες. Ελπίζουμε τελικά να καταλήξουμε σε εταιρικέ σχέσεις με τις δύο αυτές χώρες ε, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ετοιμάζουμε επίσης και το διάλογο στις 12 Δεκεμβρίου με την Ιορδανία για τη μετανάστευση, κινητικότητα και ασφάλεια και θα ξεκινήσουμε και με τη Λιβύη και την Αίγυπτο σχετικές διαπραγματεύσεις όταν οριμάσουν οι προϋποθέσεις. Ό,τι αφορά την ανατολική περιοχή, Έχουμε ξεκινήσει με την Τουρκία συμφωνίες ε, για την επανιστοχή. Βέβαια η τουρκική πλευρά ε, περιμένει ε, την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής για απελευθέρωση των θεωρήσεων ως απαραίτητη προϋπόθεση για να, υποβληθεί, για να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Θα υποβάλω αυτόν τον οδικό χάρτη, γίνονται έντονες συζητήσεις με τα κράτη-μέλη και ευελπιστούμε ότι θα ετοιμάσουμε τον οδικό χάρτη για να ξεκινήσουμε το διάλογο για την απελευθέρωση των θεωρήσεων το συντομότερο δυνατό. Επίση, θα υποβάλουμε και ένα κατάλογο με πρωτοβουλίε που θα ενταχθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασία με την Τουρκία για θέματα δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διάλογο για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, που ενδιαφέρει πολλού από εσά. Για τη δημοκρατία τη Μολδαβία έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη νομοθετική φάση και η Μολδαβία περνάει τώρα στη δεύτερη νομοθετική φάση. Για την Ουκρανία παραμένουν κάποιες εκκρεμότητες στο πλαίσιο της πάταξης των διακρίσεων και της διαφθοράς. Δεν ε, έχει ε, φέρει η Ουκρανία το, την νομοθεσία της στο απαραίτητο επίπεδο και στα βιομετρικά στοιχεία επίσης αναμένεται πρόοδος. Σε ό,τι αφορά τη Γεωργία έχει ξεκινήσει ο διάλογος από τον Ιούνιο και η νέα κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα αυτό το θέμα. Ο Ολοκληρώνουμε το σχέδιο δράση για την απελευθέρωση των θεωρήσεων και ευελπιστούμε ότι θα ξεκινήσουν όσον όπου και οι συζητήσει στο Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, έχουμε εφαρμόσει κάποια κοινά βήματα που είχαμε συμφωνήσει από πέρυσι το Δεκέμβριο. Είναι σημαντικό το θέμα από πολιτική πλευρά για τη Ρωσία. Θέλουμε όμω πρόοδο και επί τη ουσία, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό θα εξαρτήσει την ταχύτητα των εξελίσεων. Σε ό,τι αφορά ε, τι θεωρήσει. καταλήξαμε σε πολιτική συμφωνία για ένα νέο μηχανισμό αναστολή πριν από αρκετό καιρό. Αλλά λυπάμαι γιατί δεν καταφέραμε τελικά να βρούμε ε, ε, ένα νομικό συνδυασμό για τον, μηχανισμό, για τον αναθεωρημένο μηχανισμό αμοιβαιότητα. Θέλουμε έναν πιο αποτελεσματικό μηχανισμό αμοιβαιότητα. φυσικά με σεβασμό των διοργανικών συμφωνιών που προβλέπουν και συμφωνίε. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι θεμελιώδη σημασία αν θέλουμε ένα σύστημα θεωρήσεων αδιάβλητο, που θα εξασφαλίζει ίση μεταχείριση των ε, πολιτών τη ευρωπαϊκή Ένωση από εταίρου μα των τρίτων χωρών. Φυσικά οι θεωρήσει θα είναι προτεραιότητα και του χρόνου. Πριν από τρει εβδομάδες υπέβαλα μαζί με τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη τη στρατηγική ανακοίνωση για το πώ η πολιτική θεωρήσεων ε, μπορεί να συμβάλλει ε, σε ό,τι αφορά ε, την δημιουργία πολλών εκατομμύρων θέσεων απασχόληση, γιατί ο τουρισμό είναι σημαντική πηγή πλούτου και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα του κανόνε μα και να διευκολύνουμε πιο εύκολη είσοδο ε, των ε, ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτελεσματική ταυτόχρονα διαχείριση και των συνόρων μα. Γιατί μερικέ φορέ δεν θα πρέπει να αποτρέπονται τουρίστε να έρθουν στην Ευρώπη γιατί θα είναι δύσκολο να αποκτήσουν θεωρήσει. Θέλουμε κοινού κανόνε και να του αναθεωρήσουμε εφόσον επιδέχονται περισσότερο αναπλουστεύσεων. Καταργήθηκαν υποχρεώσεις θεωρήσεων για υπηκόους τρίτων χωρών που δεν δημιουργούν κίνδυνος από άποψη ε, μετανάστευσης και ασφάλειας και έχουμε ε, ένα κατάλογο ε, με, για 16 μικρά νησιωτικά κράτη της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Όλα αυτά φυσικά διευκολύνουν και τις ε, διαπροσωπικές επαφές, αλλά ε, βελτιώνουν και την οικονομική κατάσταση, γιατί οι πολιτικές εσωτερικών υποθέσεων και αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και συντόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Και μάλιστα η μεταφορά, η απόσπαση εργαζομένων, οι ε, αποσπάσεις εντός των εταιριών θα πρέπει να καλύψουν κάποια κενά στην αγορά εργασίας και να προστατεύσουν φυσικά τους εργαζομένους από τις καταχρήσεις. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να σημειωθεί πρόοδος λοιπόν στα δύο αυτά τα θέματα και προσβλέπω στην έναρξη του τριμερούς διαλόγου για το ICT με ένα πραγματικά ε, αποτελεσματικό σχέδιο κινητικότητας και να ξεκινήσουμε και για τους αποσπασμένους και τους εποχιακούς εργαζομένους της εργασίας. Χρειαζόμαστε να προσελκύσουμε και φοιτητέ και ερευνητέ όσον αφορά τον ανταγωνισμό και θέλουμε να αναθεωρήσουμε και την οδηγία για να μπορέσουμε να εντάξουμε και του κανόνε για του ερευνητέ και του φοιτητέ που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στου γενικού κανόνε υποστήριξη την οικονομία σημαίνει και να την προστατεύουμε από το οργανωμένο έγκλημα συγκεκριμένα και από το έγκλημα γενικότερα. Του χρόνου θα παρουσιάσουμε την πρώτη έκθεση κατά πολλές διαφθοράς που θα είναι τακτική με συστάσεις για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά και αυτές οι εκθάσεις ελπίζουμε ότι θα είναι ένα σημαντικότατο εργαλείο για να προσελκύσει τα μέσα των ΜΜΕ και των πολιτικών σε τομεί όπου οι προσπάθειε για την καταπολέμηση διαφθορά συστερούν και ξέρουμε ότι καμία χώρα δυστυχώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ελεύθερη από τη διαφθορά. Βέβαια η καταπολέμηση του εγκλήματος ε, δεν ε, αφορά μόνο την προστασία της νόμιμης οικονομίας, αφορά την προστασία της, των πολιτών από το έγκλημα, έχει και την ανθρώπινη διάσταση. Είμαι πολύ υπερήφανη που κάναμε βήματα τα τελευταία χρόνια στις προσπάθειες που καταβάλαμε όσον αφορά το εμπόριο ανθρώπων. Είναι ένα σημαντική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι ένα φρικτό διαδεδομένο έγκλημα και δεν ε, έπρεπε να υπάρχει το 2012. Η οδηγία κατά πολέμηση του εμπορίου ανθρώπων εφαρμόζεται σε όλο και περισσότερε χώρε και θα πρέπει μέχρι τον Απρίλιο του χρόνου να έχει πλήρω εφαρμοστεί. Και έχουμε στρατηγική όσον αφορά την καταπολέμηση του εμπορίου ανθρώπων ε, που έγινε θερμό ευπρόσδεκτο από το Κοινοβούλιο, από τα κράτη-μέλη και από άλλου εμπλεκόμενου φορεί. Τον Ιανουάριο θα εγγενιάσουμε το κέντρο καταπολέμησης του ε, εγκλήματο του κυβερνοχώρου στην Europol θα είναι εστιακό σημείο για την κοπτολέμηση των ε, εγκλημάτων του κυβερνοχώρου και είναι κρίμα που η οδηγία για τον κυβερνοχώρο δεν έχει οθετηθεί ακόμα, δοθέντω ότι καταλήξαμε σε καλό συμβιβασμό πριν από το καλοκαίρι. Ε, ολοκληρώνω με Ευρωπαϊκή Στατική Ασφαλεία του κυβερνοχώρου με την Αντιπρόεδρο Άστον βέβαια και εκεί θα δείξουμε ότι η ελευθερία και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν αποκλείουν το ένα το άλλο την επόμενη Τετάρτη μας, σαν Γενική Εισαγγελέα θα ξεκινήσω την Παγκόσμια Συμμαχία κατά τη σεξουαλική εκμεταλλεύσεω των παιδιών στο διαδίκτυο και προσβλέπω στη συμμετοχή την ευρεία Εθνικών Υπουργών και Μελών Κοινοβουλίου σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί διεθνώ και από σήμερα ήδη 46 χώρε στον κόσμο έχουν προσυπογράψει αυτή την ε, πρωτοβουλία. Γνωρίζω ότι επίσης έχουμε σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την οδηγία της κατασχέσης. Η κυρία Μακοβέη εργάζεται σκληρά πάνω σε αυτό και όλη η Επιτροπή ΚΡΙΜ για την κατάσχεση των προϊόντων εγκλήματο και προσβλέπουμε στι συστάσεις που θα μας κάνει η αρμόδια Επιτροπή για περαιτέρω βήματα που θα πρέπει να γίνουν. Τώρα όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Χαίρομαι όλους ιδιαίτερος που στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα θετήσατε την νομοθεσία για τις πρόδρομες ουσίες για τα εκρηκτικά που ήθελα ένα τεράστιο βήμα πρόοδου και προστασία των πολιτών του χρόνου. Επίσης θα ετοιμάζουμε νέα ανακοίνωση για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα όπλα, τα πυροβόλα κυρίως για να εμποδίσουμε το εμπόριο αυτών των όπλων και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια γενική πολιτική πακέτα για χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά, πυρηνικά υλικά, εκνευτικέ ύλε. Άρα θέλουμε κοινέ προσπάθειε συντονισμένε μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Όπω γνωρίζετε, επίση επιταχύνουμε το έργο μα στην αντιμετώπιση των βασικών αιτίων για, την, για, τις, για τον βίο, ριζοσπαστικές θέσεις. Είναι προσέγγιση που ακολουθήσαμε και στο δίκτυο για την ευαισθητοποίηση για το θέμα αυτών των κρυφνών θέσεων. Υπάρχουν πολλέ ομάδε που το επεξεργάζονται το θέμα και θα γίνει ένα συμπόσιο υψηλού επίπεδου τέλο Ιανουαρίου με συμμετοχή ε, εμπειρογνωμόνων και υπουργών και εκπροσώπων υπουργών. Συνεχίζουμε τι συνομιλίε με, το, με τον Καναδά για την, ε, μια συμφωνία για τα όπλα. Σημειώσαμε κάποια πρόοδο. Αλλά έχω απογοητευτεί, δεν προχωρήσαμε όσο γρήγορα θα ήθελα για να πετύχουμε ένα αποδεκτό αποτέλεσμα Ελπίζω να κάνουμε, να κάνουμε και πρόοδο και για το θέμα το, του PNR για, τις, για τους επιβάτες, επιβατών με τον Καναδά. Ε, μιλήσαμε πολύ όσον αφορά το πρόγραμμα των Αμερικανών Ασφαλές θύσεις για τη μεταφορά δεδομένων. Έστειλα μια επιστολή, αλλά δάπτω με τις ευκαιρίες να πω ότι αυτό δεν εμπίπτει στη Συμφωνία PNR Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είπα, όπως γνωρίζετε πολύ, ανήκει στο ευρύτερο θέμα των στοιχείων API, των βασικών στοιχείων που περιέχονται σε κάθε διαβατήριο επιβάτου. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημασία που έχει αυτό το θέμα και το εξετάζουμε τώρα εντελεχώ. Αυξάνεται η ανάγκη να κάνουμε περισσότερα, διότι οι περισσότερες τρίτες χώρε χρησιμοποιούν τα στοιχεία API, 32 τρίτες χώρε συλλέγουν στοιχεία και άλλες 25 σχεδιάζουν να τα συλλέξουν πολύ σύντομα και όλα τα κράτη-μέλη συλλέγουν στοιχεία API σύμφωνα με τη σχετική οδηγία. Οπότε προκύπτει ανάγκη εξέβρεση λύση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε όμω επίση να εξασφαλίζουμε ότι υπάρχει συνοχή με το διεθνέ δίκαιο και το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο. Καταλαβαίνω πολλέ από τι ανησυχίε που εκφράσατε. Το εξετάζουμε το θέμα ε, διπερισιακά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εμπειρογνώμονε και θα σα ενημερώνω θα σε ενημερώσω σύντομα σχετικά με την πρόοδο του τομέα αυτού και τέλος κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι είχαμε προτάσεις για νέο καταστατικό για την Ευρωπόλ και μεταρρυθμίσεις της ΕΠΟΛ ε, και το καταστατικό. έχουμε περικοπές προβλέψει σε παγκόσμιο επίπεδο στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, πολιτικό πλαίσιο και θέλουμε να δούμε πώς θα ε, κάνουμε καλύτερη κατανομή του προσωπικού. Το εξήγησε ο κ. πριν από κάποιες μέρες. Θέλουμε να συγχωνεύσουμε Ευρωπόλ και ΣΕΠΟΛ για τις περικοπές αυτές. Αυτό θα συνεπιφέρει σημαντικές οικονομίες όσον αφορά το κόστος των διαφόρων γραφείων και υπηρεσιών και θα έχουμε αποτελεσματικότατο πρόγραμμα κατάρτισης, διότι δεν προτιθέμεθα να υποβαθμίσουμε την κατάρτιση αστυνομικών, αντιθέτως μάλιστα, θέλουμε να έχουμε πολύ φιλόδοξα επίπεδα εκπαίδευση αστυνομικών και θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την προσπάθεια. Δεν έχουν ληφθεί ακόμα αποφάσεις, αλλά ήθελα να ξέρετε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις όσον αφορά την πρόταση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, θέλαμε να απλουστεύσουμε τη χρηματοδότηση των θεμάτων εσωτερικών και θέλαμε να δώσουμε χώρο και στην εξωτερική διάσταση των εργασιών. Πετύχαμε πρόοδο εδώ και στο Συμβούλιο. Βεβαίω η πρόοδο εξαρτάται από το γενικό ύψο του προπολογισμού και όπω όλοι γνωρίζετε δεν υπήρξε συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτό το Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε λοιπόν ότι ο προπολογισμό στο θέμα αυτό θα επιληθεί σύντομα, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε το διάλογο για την πολιτική αυτή με κάθε κράτο μέλο σε ευθέτω χρόνο. Είναι σημαντικό κομμάτι του νέου συστήματο θέσει προτεραιοτήτων για τη χρηματοδότηση. Εδώ ελπίζω κύριε Πρόεδρε να κάλυψα πολλά ζητήματα ενδιαφέροντο, βεβαίω όχι όλα, αλλά είμαι έτοιμη να ακούσω σχόλια και ερωτήσει, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. Thank you. Ευχαριστώ, Επίτροπε Μάλμστρομ. Καλό σας απόγευμα σε όλους. Καθυστέρησα σε μποτιλιάρισμα και μου πήρε πάνω από μία ώρα για να έρθω από το αεροδρόμιο εδώ. Λόγω των διαδηλώσεων με τρακτέρ κατά, η διαδήλωση είναι κατά των προοπτικών της κοινή αγροτικής πολιτικής. Αυτό όμως είναι μια εξήγηση μόνο για να δικαιολογηθώ γιατί δεν ήμουν εδώ από το πρώτο λεπτό. Ευχαριστώ που ήρθατε, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας σε σχέση με τις εξελίξεις και την εφαρμογή των προοπτικών που ετέθησαν όταν εγκρίναμε το ψήφισμα για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και την ε, ενδιάμεση εξέταση, επανεξέταση. Τώρα προσεγγίζουμε το τελικό χρόνο αυτού του προγράμματος 2009-2014. Πριν δώσω το λόγο στα μέλη που θέλουν να συμβάλλουν, έχω έναν κατάλογο εδώ, ως αρμόδιος εισηγητής ε, για αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας που αποφασίστηκε από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα ήθελα να πω δύο λόγια λοιπόν σε σχέση με την προοπτική των εργασιών μας. Κάναμε μία συνάντηση την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Συγκάλεσα την συνάντηση με τους Κιώδης και τους συντονιστές της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για ανταλλαγή απόψεων και για να διαβεβαιώσω ότι ως εισηγητής θα συνεργαστώ στενά με τους ε, σκιώδεις εισηγητές για να ε, γίνει αυτή η ενδιάμεση επανεξέταση. Θα ήθελα να θυμίσω ότι μια εβδομάδα από τώρα έχουμε την πρώτη επέτειο Τη συνθήκη της Λισαβόνας που ετέθησε ισχύ το 1η Δεκεμβρίου του 2009. Θα είναι δηλαδή η επέτειος των τριών ετών τώρα, σε λίγες μέρες. Και αυτό είναι μια ευκαιρία για να δούμε λίγο πώς προχώρησαν οι εξελίξεις Γνωρίζουμε όλοι ότι έχει γίνει πρόοδος και βεβαίως αναγνωρίζουμε και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Κομισιόν, ιδιαίτερα στον τομέα του ασύλου, και είμαστε βέβαιοι ότι σύντομα θα, θα ολοκληρωθεί το έργο εκεί, αλλά έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε επίσης σε άλλους τομείς που δεν έχουν τόσο θετικές ε, δεν ήταν τόσο θετική η επανεξέταση για την Europol, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ζήτησε πρόταση πριν από την, ε, ε, το, 2010, οπότε έχει καθυστερήσει το προγραμματικό μας έργο και εξακολουθεί να αναβάλλεται, αυτό είναι μια λεπτομέρεια ίσως, αλλά αυτό σημαίνει ότι τρία χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, η Europol εξακολουθεί να λειτουργεί όπως λειτουργούσε πριν τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Και αν η πρόταση δεν υποβληθεί σύντομα, ε, δεν θα προλάβουμε να κάνουμε τη δουλειά που πρέπει λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 θα είναι το τελευταίο επιχειρησιακό έτος εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις πρώτες μήνες του 2014 θα είμαστε μπροστά στις ευρωεκλογές και θα επικεντρωθούμε στην σημασία της ημέρας αυτής και τον πολιτικό ανταγωνισμό που κρύβεται πίσω από τις εκλογές. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το θυμίσουμε να μην χαθεί ούτε λεπτό, ούτε δευτερόλεπτο από το χρόνο που έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας. Και χρειάζεται επακριβή σχεδιασμό των προτάσεων από την DG Home και το δικό, εσωτερικών και το δικό σας χαρτοφυλάκιο. Δεύτερον, έλεγχος της εφαρμογής, του κεφαλαίου της εφαρμογής υλοποίησης. Το πρόγραμμα της ε, Στοκόλμης λέει ότι θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να προσέξουμε ιδιαίτερα την πλήρη και αποτελεσματική ε, εφαρμογή της ε, επιβολής του νόμου. Οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να ωφελούνται από το χώρο δικαιοσύνης, ελευθερίας, ασφάλειας και γι' αυτό θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι πολιτικές της Ένωσης θα εφαρμόζονται σωστά από τα κράτη-μέλη. Συζητούμε λοιπόν το πακέτο διακυβέρνησης του Σέγγεν. Ε, ακούσαμε συχνά από τα κράτη-μέλη να λένε ότι όλα είναι εντάξει αφού ακόμα δεν έχει, δεν έχει αρχίσει η Κομισιόν διαδικασίες επί παραβάση, αλλά πρέπει να μπούμε λίγο πιο βαθιά στο θέμα αυτό, γιατί το πακέτο διακυβέρνησης του Σένιεν πραγματικά ε, πρέπει να εφαρμοστεί σωστά. Και η έλλειψη της ε, διαδικασίας επί παραβάση είναι αρκετά καλά νέα, γιατί πρέπει να εμβαθύνουμε εδώ. Τέλος, θα ήθελα να πω κάτι σημαντικό για τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων και την πλήρη ένταξη βέβαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Κοινοβουλίου στο έργο αυτό. Η συνθήκη της Λισαβόνας ζητεί πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ανάπτυξη στρατηγικών και προγραμμάτων και οι στρατηγικές ε, αποφάσεις θα γίνονται με βάση την νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει δημόσια συζήτηση ε, και διαβουλεύσεις στα θέματα που διακυβεύονται θα γίνει μια συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια για την αξιολόγηση του προγράμματος της Στοκχόλμης την Άνοιξη τον επόμενο χρόνο. Ε, αρκετά ε, θέματα αφορούν την ε, συγκεκριμένη διάταξη της συνθήκης της Λισαβόνας, αλλά η συνθήκη της Λισαβόνας στο πρωτόκολλο 36 ε, αναφέρει ένα πενταετές πρόγραμμα για ε, ε, περάσει το κεκτημένο του πρώην τρίτου πυλώνα στο καθεστώς της Λισαβόνας. Δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε, πρέπει να κινηθούμε στοχευμένα για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και υπ' αυτή την έννοια σας διαβεβαιώνω ότι συνεχίζουμε να είμαστε απόλυτα έτοιμοι να συνεργαστούμε για όλα αυτά με την Κομισιόν. Μετά από αυτό, αφού αναφέρθηκα στο σκοπό της έκθεσης που συζητούμε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στα μέλη που ζήτησαν, αρχίζοντας από τον κύριο Κοέλιο. Thank you so much, Chairman. Um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Ευχαριστώ τη Σισίλια Μάλθον για τα στοιχεία που έδωσε στην Επιτροπή μας. Και θέλω να ρωτήσω εξ από τον κύριο Ντεμέρα που δεν μπορεί να είναι εδώ, πότε η Κομισιόν θα στείλει στο Κοινοβούλιο τις προτάσεις για την Europol. Είναι συγκεκριμένο το ερώτημα. Η Σεσίλια Μάλμστρο μίλησε για το SIS, το Schengen Information System. Δεν θα ξανακάνουμε τη συζήτηση που είχαμε στο Στρασβούργο. Αλλά Μόνο μια μικρή ερώτηση. Ελπίζομαι ότι δεν θα τροποποιηθεί το πρόγραμμα της νέας Κομισιόν από όλα αυτά. Ελπίζω ότι μιλάμε για μια τρίμηνη μόνο παρα... αναβολή. Αλλά υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα σε ορισμένες χώρες Σουηδία, Νορβηγία, εντάξει δεν είναι η τελευταία κράτος μέλος, αλλά είναι τέρος στο Σέγγεν και Φιλανδία. Υπάρχουν χώρες λοιπόν βόρειες που έχουν προβλήματα με τη βάση δεδομένων, με, με τα διαβατήρια που έχουν εκεί και ελπίζω ότι δεν θα ανακύψουν καινούργια προβλήματα στις χώρες αυτές. Και δεν ξέρω, ρωτώ την ε, Σεσίλια Μάλμστρομ αν μπορεί να μας ενημερώσει. Τέλος, ε, η Επίτροπος δεν θα είναι στο δεύτερο μέρος της συζήτησης για τη διακυβέρνηση του Σέγγεν, θα είναι ο κύριος Μοσχοβησή, αλλά είναι πολιτικό το ερώτημα που θέλω να θέσω στη Σεσίλια Μάλμστρομ και αφορά την αποδοτικότητα της νέας διακυβέρνησης του Σέγγεν. Στην τελευταία συνεδρίαση και τριμερή διάλογο που είχαμε και με Συμβούλιο και με Κομισιόν, αντιληφθήκαμε ότι το Συμβούλιο δεν θέλει να ληφθεί απόφαση ε, για την κατάργηση των συνοριακών ελέγχων. Δηλαδή όλο το οικοδόμημα που είχαμε προβλέψει, δηλαδή ότι όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα μπορούμε να ε, ε, ε τα λύνουμε και να αποφασίζει ολόκληρη η περιοχή Σένιν για του συνοριακούς ελέγχου. και το θέμα ήταν αν θα λάμβανε την απόφαση Κομισιόν ή το Συμβούλιο. Τα τελευταία νέα είναι ότι το Συμβούλιο δεν θέλει καμία απόφαση. Ούτε από την Κομισιόν, ούτε από το Συμβούλιο. Από ό,τι φαίνεται γιατί τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να λαμβάνονται αποφάσεις για τα σύνορά τους. Ε, είναι στο χέρι των κρατών μελών να αποφασίζουν. Οπότε μένουμε εκεί που είμαστε. Το πολιτικό ερώτημα προς την Επίτροπο είναι αν το Συμβούλιο δεν ε, είναι διατεθειμένο να δώσει λύση την ασφάλεια του χώρου Σέγγεν, Υπάρχει λόγος να συνεχίζονται διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία που θα διατηρεί τους ίδιους κανόνες που έχουμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζίμπελ. Κυρία... Όχι, δεν ζήτησε το λόγο. Ο κύριος ε, Έλσιου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ θερμά για την ε, ομιλία σας, για την παρουσίαση που μας κάνατε και θα ήθελα να σας εκφράσω τη χαρά μου για το γεγονός ε, της επίσκεψής σας, αλλά λυπούμε ταυτόχρονα για την απουσία σας από την τελευταία ολομέλεια του Στρασβούργου. Γιατί τότε μας ε, χρειάζονταν αυτές οι πληροφορίες για το πρόγραμμα πληροφοριών ε, Σέγγεν για το ΣΥΣ 2. Όπως ε, είπε και ο Πρόεδρος ε, και ο κύριος Κοέλιο, θα θέλαμε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για την ε, επίσκεψή σας στη Φιλανδία και τι προέκυψε από την επίσκεψη εκείνη. Θα προκαλέσει καθυστερήσεις η Φιλανδία σε όλη αυτή την προσπάθεια μετάβαση από το ΣΥΣ 1 στο ΣΥΣ 2 δεδομένη της ε, μεγάλη χρονοτριβή που ήδη διαπιστώσαμε στη μετάβαση αυτή. Και σε ό,τι αφορά το πακέτο διακυβέρνηση τη ζώνη Σέγγεν, που αποτελεί ένα ε, σημαντικό θεμελιώδες τμήμα του προγράμματος της Στοκχόλμης. Όπως είπε και ο κύριος Κοέλιο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων ε, κατέληξαν σε αδιέξοδο. Και δεδομένων των μεγάλων διαφορών και της μεγάλης διάστασης απόψεων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι για την έκβαση αυτών των συζητήσεων. Οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οπωσδήποτε να παίξει κεντρικό ρόλο στη νέα πρόταση. Και γνωρίζουμε ε, γιατί το Συμβούλιο διαφωνεί κάθετα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαδραματίσει ένα θεμελιώδη ρόλο και να απεμπλέξει το διέξοδο αυτό και την αποτελμάτωση που διαπιστώνουμε στις συζητήσεις για το πακέτο διακυβέρνησης Σέγγεν. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που παραλείψατε εσείς στην παρουσίασή σας. Τι γίνεται με το νέο πακέτο για τα smart waters, γιατί περιμένουμε ε, να υποβληθεί αυτό το πακέτο, το, το πακέτο των ε, smart borders, διορθώνει μιλητή, των ε, έξυπνων συνόρων, να υποβληθεί το συντομότερο δυνατό πριν το τέλη ίσως του 2012. Και επίσης περιμένουμε σημαντικές περικοπές κατά δύο δις το πακέτο αυτού με τόσο δραστικές περικοπές θα μπορέσει παρόλα αυτά να επιβιώσει αυτό το πακέτο για τα έξυπνα σύνορα. Και τέλος, ένα άλλο θέμα που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλέ αφορά φυσικά την πλήρη ένταξη της Ρουμανία και Βουλγαρίας στο χώρο Σέγγεν. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ε, προσωπική σας ε, θέση υπέρ της πλήρους ένταξη των δύο χωρών. Να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη που μας παρήχατε και να σας συγχαρώ. Όπως διαπιστώσατε με το επεισόδιο αυτό που είχαμε για το ΣΥΣ2, η Ρουμανία και η Βουλγαρία πληρούν ήδη όλα τα κριτήρια για να ενταχθούν πλήρως στη ζώνη Σέγγεν, στο χώρο Σέγγεν. Και επιπλέον οι δύο αυτές χώρες είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένες από μερικές παλιές χώρες του χώρου Σέγγεν. Είναι έτοιμες να περάσουν χωρίς κανένα πρόβλημα στο ΣΥΣ2. Φαίνεται ότι εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά λοιπόν. Η κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επίτροπο που ήρθε σήμερα στην ε, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για να μας κάνει αυτή την ενημέρωση θα ήθελα να εκφράσω την βαθύτατη μου θλίψη για το γεγονός ότι το πακέτο και του ασύλου και της μετανάστευσης υποβάλλονται σε μια εποχή που δυστυχώς έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχοντας λοιπόν αυτό το θέμα υπόψη και τις αντιστάσεις του Συμβουλίου για κάποιες πτυχές αυτού του πακέτου, δεν μπορούμε να παρά να διαπιστώσουμε ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Και ελπίζουμε ότι σε τελική ανάλυση θα έχουμε τουλάχιστον κάποιες ε, ελάχιστες προδιαγραφές. Παρά είναι βέβαια ε, ελάχιστες κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ λίγο φιλόδοξος αυτός ο στόχος, αλλά φαίνεται ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει πολύ περισσότερους τομείς από ότι ε, μόνο την οικονομία. Έχει αγγίξει πραγματικά τις ψυχές των ανθρώπων πολύ πιο βαθιά. Και καλό βέβαια να λέμε για το εθνικό συμφέρον, αλλά μερικές φορές ε, ο λαϊκισμός βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτή την ε, αγκίστρωση, σε αυτό το εθνικό συμφέρον. Τώρα και έχω και μια συγκεκριμένη ερώτηση από τον συνάδελφο Βίλντεν που ήταν και επικεφαλής της αντιπροσωπείας που μετέβη στην Ελλάδα πριν από λίγες εβδομάδες. Ο Γιάνν Μούλντερ είναι ένας πολύ λογικός άνθρωπος, συνετός, ισορροπημένος και μετράει τα λόγια του και τις εκτιμήσεις του. Όταν λοιπόν ο Γιάνν Μούλντερ ε, δηλώνει ότι συναντήθηκε με αξιωματούχους της αστυνομίας, με ανθρώπους ιδιαίτερα αφοσιωμένους, ε, εγώ τον πιστεύω γιατί γνωρίζω πώς ε, παρουσιάζει με λογική και ακρίβεια την κατάσταση. Όταν όμως ο ίδιος ο Γιάνν Μίλντερ λέει ότι σε μερικά κέντρα, ε, στο Βίνι και στο Ελληνικό, η κατάσταση ήταν αποτροπιαστική και πάλι όταν δηλώνει κάτι τέτοιο Γιάνν Μιούλτερ εγώ τον πιστεύω. Η κατάσταση ήταν πραγματικά τρομακτική. Και μάλιστα σε αυτά τα δύο κέντρα και εσείς πήγατε ένα μήνα πριν τον Γιάν Μίλντερ και είπατε ότι θα ακούσατε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα κλείσουν αυτά τα κέντρα. Ο Γιάν Μίλντερ τώρα άκουσε ότι τα κέντρα αυτά θα κλείσουν τον Απρίλιο. Οπότε η πρώτη ερώτηση είναι τι συνέβη τελικά. Γιατί και ο Γιάν Μίλντερ με την αντιπροσωπεία πήγε σε ένα κέντρο κοντά στην Αθήνα και μάλιστα εκεί υπήρχαν ακόμη ε, ελεύθερες θέσεις. Υπήρχε χώρος για, να υποδοχή, για, και περισσό, για υποδοχή περισσότερων, οπότε από διοικητική άποψη κάτι θα μπορούσε να γίνει. Και ένα άλλο ερώτημα, μια άλλη απορία που προέκυψε από την επίσκεψη αυτή είναι ποια είναι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή την ε, δυνατότητα να βοηθούν ε, και οικονομικά οι ελληνικές αρχές για να δημιουργήσουν και άλλα κέντρα για να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους ε, να ξεφύγουν από αυτή τη δινή κατάσταση. Αλλά δυστυχώς υπάρχει έλλειμμα αλληλεγγύης όπως είπα και προηγουμένως. Και φυσικά δεν θα μπορούσα να μην ασχοληθώ και με το ζήτημα του Σέγγεν. Ίσως θα μπορούσα να αναδιατυπώσω κάπως ε, την ερώτηση και να προσπαθήσω να καταλάβω ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε για το Σέγγεν. Τώρα γίνονται οι διαπραγματεύσεις ε, των δύο τμήματων αυτού του πακέτου. Για μας ήταν από την αρχή σαφές ότι ενώ δεν θέλαμε να έχουμε μια νέα δυνατότητα για επανεισαγωγή του, του ελέγχου στα σύνορα, ήμασταν απόλυτα ανοιχτοί ως προς ένα μηχανισμό που θα βοηθούσε μια χώρα που είτε δεν δύναται, είτε δεν επιθυμεί να ελέγξει τα εσωτερικά της ε, σύνορα, να τη βοηθήσουμε. Και αν ε, αυτή η προσπάθεια ήταν ατελέσφορη, θα ζητούσαμε από τις άλλες χώρες να επαναφέρουν τα, τους ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα και θέλαμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο να τον διαδραματίσει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και φάνηκε αυτό και από την ψηφοφορία, γιατί είναι φυσιολογικό ε, κάποιο ουδέτερο μέρο να λαμβάνει την απόφαση. Τώρα αυτό που μας λέει το Συμβούλιο είναι ότι μια τέτοια απόφαση, και αυτό φυσικά στηρίζεται και στην γνωμοδότηση της νομικής τους υπηρεσίας, που είναι απόρριτη και εμπιστευτική, πολύ ωραία όλα αυτά για τη διαφάνεια, λέει λοιπόν, μας είπαν τουλάχιστον ότι αυτό λέει η γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας, ότι κάτι τέτοιο θα θεωρούνταν ως τρόπο επιβολής κυρώσεων στα κράτη-μέλη. Γιατί ένα κράτος δεν θέλει να συμμορφωθεί με τις συστάσεις και τα λοιπά και τα, υπόλοιπα θέματα, τότε η επανεισαγωγή του ελέγχου στα σύνορα και η απόφαση να, υποχρεωθεί ένα κράτος να επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορα, αυτό δυναμή με κύρωση. Οπότε ούτε το Συμβούλιο, ούτε η Επιτροπή. Γιατί ήμασταν έτοιμοι να δεχτούμε μια τέτοια απόφαση ακόμη και το Συμβούλιο, αλλά φαίνεται ότι ούτε το Συμβούλιο ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνονται να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό που πρότεινε το Συμβούλιο τελικά είναι να υποβληθεί απλώ μια σύσταση. Και μάλιστα όχι στην υπεύθυνη χώρα, αλλά στι γειτονικέ χώρε, στι όμορε τη χώρα. Οπότε το θέμα δεν είναι ε, τι είναι το χειρότερο να σταματήσουμε τις διαπραγματεύσεις, γιατί μετά από ένα μισή χρόνο εδώ έχουμε φτάσει μόνο. Θα ήθελα όμως να ακούσω τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πού είναι διατεθειμένη να φτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι υποχωρήσει να κάνει και ποιες προτάσεις του Συμβουλίου να αποδεχθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και Βέμπερ. Επόμενος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε διεξοδικότατη παρουσίαση της ε, πρόοδου στο πρόγραμμα Στοκχόλμης. Είναι πολύ σημαντικό να αξιολογήσουμε το πώς εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, να δούμε τι χρειάζεται ακόμα να γίνει. Δεύτερον, να προετοιμαστούμε για το επόμενο πρόγραμμα. Για να κινηθούμε σωστά, λαμβάνοντας υπόψη στους πολίτες, χρειάζεται διαφάνεια στην διαμόρφωση πολιτικής. Για τούτο, σας ζητούμε να μας στείλετε συγκριτικό πίνακα που θα εμπεριέχει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με σχέδιο δράσης για τη Στοκόλμη, τις προτάσεις που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα αναμοθετήματα που έχουν υιοθετηθεί. Αυτό θα μας βοηθήσει να σχηματίσουμε μια εικόνα σχετικά με την παρούσα κατάσταση. Επίτροπε, όσον αφορά τη γνώση της θέσης μας, γιατί υπάρχουν οι πίνακες που βαθμολόγηση που υπήρχαν κατά το παρελθόν δεν υπάρχουν πλέον. Είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντο το θέμα για μένα. Σας ερωτώ, τι σημαίνει όσον αφορά την αλληλεγγύη στον τομέα του ασύλου. Έχουμε την εντύπωση ότι έχουν κολλήσει τα πράγματα. Βλέπουμε εκρήξεις βίας και αυξανόμενο ρατσισμό και ξενοφοβία. Πότε σχεδιάζετε να εφαρμόσετε τα όσα ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του Πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγησή σας και πότε θα υποβάλλετε πρόταση για μηχανισμούς ε, μετεγκατάστασης. Και άλλη ερώτηση αν επιτρέπετε. Η ανακοίνωσή σας για νέες προσεγγίσεις για πρόσφαση σε διαδικασίες ασύλου για τις χώρες διέλευσης πότε θα υποβληθεί και το πλαίσιο για μεταφορά προστασίας δικαιούχων διεθνούς προστασίας και αμοιβαία αναγνώριση ε, αποφάσεων για το άσυλο. Αυτά πότε θα κινηθούν αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί Επίτροπε, σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για την σημερινή σας παρουσίαση. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω. Δημοσία. Εκφράζω την εκτίμησή μας για τις προσπάθειες που καταβάλατε για να υποστηρίξετε τη χώρα μας στο τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου. Και μάλιστα το τελευταίο τετράμινο-πεντάμινο είχα ερώτηση γενικότερου περιεχομένου, αλλά μετά τις ερωτήσεις κυρίας Βέμπερ θέλω να πω ότι μια αντιπροσωπεία πήγε στην Ελλάδα εδώ και ένα μήνα μέλη της Επιτροπής ε, Ελευθεριών επισκέφτηκαν κέντρα στην Αθήνα έγιναν πολλές συνεδριάσεις και συναντήσεις. Συμπέρασμα μετά την αποστολή είναι ότι αυτή την περίοδο δίνει αποτελέσματα, πετυχαίνει αποτελέσματα η Ελλάδα. Ελπίζω να αποκομίσετε την ίδια εντύπωση όταν, πριν από, όταν την Ελλάδα, δύο εβδομάδες πριν επισκεφτούμε εμείς την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο το ότι είχαμε την υποστήριξη Ευρωπαϊκή Επιτροπής έγινε τροποποίηση των πόρων για καλύτερη απορρόφηση της χρηματοδότησης και να χρησιμοποιήσουμε τη Frontex και άλλα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η στήριξη και βοηθά την, ε, τις ελληνικές προσπάθειες και στους επόμενους μήνες. Στην αντιπροσωπή αυτή, στην επίσκεψη, είχαμε τη δυνατότητα να δούμε και τα προβλήματα. Επισκεφθήκαμε δύο κέντρα ένα στον Εύρο και ένα στο Ελληνικό, στην Αθήνα. Εκεί πράγματι υπάρχουν προβλήματα. Θα σας ενημέρωσαν οι ελληνικές αρχές ε, που θα σας είπαν ότι σύντομα ευτυχώ θα κλείσουν αυτά τα κέντρα. Αυτό ήταν αίτημα όχι μόνο των συναδέλφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Δεν θέλει κοινωνία αυτά τα κέντρα. Νομίζω ότι και τα άλλα κέντρα που επισκεφθήκαμε ε, είναι σε καλή κατάσταση δημιουργούνται νέα κέντρα αυτή την περίοδο και έχει σχεδιαστεί να δημιουργηθούν και άλλα τους επόμενους μήνες για, ε, για υποδοχή ε, υπηκών χωρών, πρώτη υποδοχή. Ερώτηση μετά τα όσα μας είπε και ο Τερνταφυλίδης. Όταν ήρθαμε στο Κοινοβούλιο θυμάμαι ότι ένα από τα πρώτα θέματά μας ήταν το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και πάνω σε αυτό επέβαλα τις πρώτες μοτροπολογίες, εκεί αναφερόταν η αλληλεγγύη και σε σχέση με αυτή την αλληλεγγύη περιμέναμε την ανακοίνωση για τις μετεγκαταστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το, στο ψήφισμά μας βάσει τη εκθέσεω του κ. Τριανταφυλλίδη, ένα ψήφισμα που πέρασε πριν από δύο μήνες, αναφέραμε και την κλίδα κατανομής που απαιτείται για τους ετούντες ασυλώς σε εξαιρετικές περιστάσεις για χώρες που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πίεση. Έχουμε κάποιες ειδήσει όσον αφορά την ε, ανακοίνωση αυτή. Πρόκειται να συμπεριλαμβάνεται και κλίδα κατανομής στην ανακοίνωση αυτή για τις μετεγκαταστάσεις. Και στην επίσκεψή μας στην Ελλάδα είδαμε κάτι που συζητάμε και εδώ. Υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότησης για την Frontex και την EASO ότι δεν, υπά, αρκετά, δεν είναι αρκετά τα χρήματα για τις κοινέ επιχειρήσεις που απαιτούνται σε πολλές περιπτώσεις. Έχετε κάτι υπόψη σας γι' αυτό. Ο διευθυντής της Frontex πρόσφατα ήρθε εδώ και είπε τα ίδια. Ζητούν περισσότερα χρήματα οι υπηρεσίες αυτές. Αναμένετε κάτι καινούριο από την πλευρά σα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκεγιόμ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση, κυρία Μάλστρομ. Όσον αφορά το πρόγραμμα, θυμάμαι πολύ καλά όταν μιλήσαμε στην αρχή για το θέμα αυτό και ψηφίσαμε το πρόγραμμα και λέγαμε ότι υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται σημαντικές πρόοδοι και λήφθησαν υπόψη οι τροπολογίες για την επίτευξη καλύτερη ισορροπία μεταξύ του σεβασμού του ατόμου και τα χέγγια για μια ασφάλεια βιώσιμη για τους πολίτες. Και βλέπουμε μετά με τον κατάλογο που μας δώσατε, που είναι αρκετά μακροσκελής και ενδεικτικό ότι έχουν δρομολογηθεί πολλά προγράμματα, μερικά από αυτά ακολουθούν καλό δρόμο, αλλά και κάποιες διατάξεις αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν αποτελμάτωση όχι απεραίτητα λόγω προβλημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ίσως να μην δίνεται η σωστή εικόνα για τα προγράμματα, δεν τόσο ιδεώδης. Και στην εφαρμογή τους τα προγράμματα δεν εφαρμόζονται σε ουδέτερη περίοδο, όλα οικονομικής κρίσης πολύ μεγάλης, που όσον αφορά τη μετανάστευση ε, έχει συνέπειες όσον αφορά τη μετακίνηση των ανθρώπων θα ήταν ενδιαφέρον αυτό να το εξετάσουμε επακριβώς, διότι νομίζω ότι η κρίση ε, όσον αφορά τις ροές σε κάποιες περιοχές έχει επιρροή και επηρεάζει η κρίση και πολύ τις αντιδράσεις των κρατών μελών. Αναφέρθηκε προηγουμένως αυτό. Όταν έχουμε οικονομικούς περιορισμούς, μιλάμε, ε, τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πολύ ακριβά και, δεν, και γι' αυτό μπλοκάρονται και δεν εφαρμόζονται αρκετά γρήγορα. Και αυτό επηρεάζει και την ελληνική. Επηρεαστήκαμε και από την Αραβική Άνοιξη και τις αποφάσεις που ελήφθησαν από κάποια κράτη-μέλη. Όμως και αυτά ε, θα συζητηθούν και θα εξεταστούν. Αναγνωρίζω τη δουλειά που έγινε. Αλλά εκφράζω τη λύπη μου για τρία πράγματα. Μπορείτε να μας απαντήσετε, να εκφράσετε απόψη πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, το θέμα της αλληλεγγύης είναι που με προβληματίζει. Σημαντικότατο θέμα, σημαντικότατο σημείο του προγράμματος Στοκχόλμης, είχαμε επιμείνει πολύ από αυτού. Φοβούμαι όμως ότι όσον αφορά την τυχή αυτή της ευθύνη αλληλεγγύης και τη συνεργασία όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση που είναι ένα από τα προγράμματα της ένα, μια από τις του προγράμματος της Στοχόλμης υπάρχουν όρια όσον αφορά την ελληνική και πόρο απέχουμε από, την, από τον ισότιμο επιμερισμό των ευθυνών. Θα ήθελα να σας ακούσω από αυτού. Δεύτερον, δεύτερον εκφράζω τη λύπη μου διότι η μεταναστευτική διάσταση στην εφαρμογή κάποιων προγραμμάτων και διατάξεων έχει μείνει κάπω πίσω. Και η πρόθεση τη ένταξη και των δικαιωμάτων των μεταναστών ακόμα είναι ο φτωχό συγγενή των κοινοτικών δράσεων. Πώ μπορούμε κατά την άποψή σα να προωθήσουμε κάποιε ιδέε, κάποιε διατάξει ούτω ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε όσον αφορά τα δικαιώματα αυτά στο μέλλον. Τρίτο σημείο που εκφράζω τη θλίψη μου και απευθύνω και έκκληση για την άποψή σα. Ε, είναι το θέμα του κοινού καθεστώτος για το άσυλο, όπως και εσείς Έχω κάθε εμπιστοσύνη στην ταχεία υλοποίηση. Ε, χρειάζεται όμως όχι μόνο ελπίδα αλλά και δουλειά πάνω σε αυτό. Θα θέλαμε ε, κάπου να καταλήξουμε κυρίως με τον λογική των τελευταίων κειμένων όσον αφορά τα διαδικαστικά θέματα να καταλήξουμε κάπου. Επίσης και ο ρόλος του Κοινοβουλίου που είναι συνομοθέτης θα πρέπει να γίνει σεβαστός και θα πρέπει να εισακουστούν τα όρια που θέτουμε οι κόκκινες γραμμές. Και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανεπάρκεια προόδου σε κάποιες διαστάσεις και όσον αφορά το, ε, αυτά τα θέματα που σας ανέφερα. Ευχαριστώ κυρία Ιντβερτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που μας ε, δώσατε αυτή την συνολική, ε, μας κάνετε αυτή τη συνολική παρουσίαση. Μιλήσατε για ασφαλείς πτήσεις. Χαίρομαι που το λέτε μετά από πάρα πολλές ερωτήσεις που τα προηγούμενα χρόνια υποβάλαμε. Χαίρομαι που επιτέλους ημερίζεστε την ανησυχία μας γιατί δεδομένα διαβιβάζονται χωρίς νομική βάση. Το έχουμε πει με την Κομισιόν πολλές φορές, το έχουμε θέσει το θέμα και περιμένουμε περιέργεια να δω τι θα κάνετε. Ε, PNR με τον Καναδά. Δεν ξέρω τι να πω. Ε, έχει γίνει πια αστείο το πράγμα. Είτε θα υπάρχει νομική βάση για τη διαβίβαση δεδομένων και δεν χρειάζεται διαπραγμάτευση, ή δεν, ή δεν υπάρχει και είμαστε σε κατάσταση παρανομίας, δεν ξέρω πόσα χρόνια τώρα, και δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζονται δυόμιση χρόνια διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία εδώ. Τρίτον, ε, κάτι που ίσω το αναφέρατε, αλλά μου διέφυγε ή δεν το αναφέρατε, δεν ξέρω. Είναι το TFTS, όπως λέγεται τώρα, που δεν μου αρέσει και πολύ όπως ξέρετε, δεν είναι μυστικό αυτό, και θα ήθελα να μου πείτε, οι προτάσεις, οι επικείμενες προτάσεις, πώς σχετίζονται με την συμφωνία SWIFT που φαίνεται να μην είναι ικανοποιητική. Και περνώ στο τέταρτο θέμα της διαφάνειας που δεν είναι ε, αυστηρά δική σας αρμοδιότητα, αλλά όχι μόνο έχουμε διαπραγματεύσεις για την επανεξέταση του κανονισμού για τη δημόσια πρόσβαση στα δεδομένα, όχι μόνο δεν κατέρευσαν, αλλά και ο τωρινός κανονισμός δεν λειτουργεί καλά. Γιατί ως κοινοβούλιο δεν μπορούμε να ασκήσουμε αποτελεσματικό έλεγχο της ε, εφαρμογής της συμφωνίας. Συμφωνήσαμε απρόθυμα να εγκρίνουμε τη συμφωνία. Μετά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια έκθεση, η σύνοψη της οποίας φαίνεται να υποδηλώνει ότι ε, σε τελευταία ανάλυση δεν ενδιαφέρεται κανείς και τα δεδομένα πάνε έτσι και λέει στους Αμερικανούς. Και η μόνη πίεση που μπορούμε να ασκήσουμε ως Κοινοβούλιο είναι να ε, ασκήσουμε πολύ στενή παρακολούθηση της συμφωνίας. Όποτε το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί σε κάτι, έχει αυτή τη μαγική φόρμουλα. Το δεχόμαστε, αλλά θα το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ. Μα πώ να το κάνουμε αυτό, αφού δεν έχουμε πρόσβαση στην πληροφόρηση. Και τέλο, και φαντάζομαι ότι θα το κατανοείτε πολύ αυτό, γιατί εσεί είσαστε μία από τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από τον κανονισμό για τη διαφάνεια. Τέλος, για την διατήρηση των δεδομένων, είμαι περίεργη να ακούσω τι θα κάνουμε σε αυτό το μέτωπο, γιατί από ό,τι κατάλαβα, δεν ε, υπήρξε πιστική απόδειξη της χρησιμότητας, για να μην πω για αναγκαιότητα της οδηγίας. Αμφισβητήθηκε σε πολλά κράτη-μέλη, έχει πάει στα δικαστήρια. Χθες ε, είδαμε πάλι μια αναφορά, αυτή τη φορά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ολλανδίας, που λέει ότι οι αστυνομικές δυνάμεις ελεύθερα κοιτάνε τα, τις βάσεις δεδομένων χωρίς να δίνουν καμία σημασία στους κανόνες. Οπότε δεν βλέπω γιατί εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε μια οδηγία η οποία δεν καταξιώθηκε, δεν απέδειξε τη χρησιμότητά της. Αντίθετα, έδειξε τα μειον, πολλά Τι συνέχεια θα δοθεί εδώ. Ευχαριστώ. Τέλος, η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν άκουσα την παρέμβασή σας, αλλά βλέπετε Ήμουνα σε μια άλλη συνεδρίαση και θα ήθελα να εκφράσω τις ανησυχίες μου όσον αφορά τα κονδύλια που δίνουν σε κάποιες φορέ κυρίως της ΕΠΟΛ, την Ευρωπόλ και την Γεροζίστ Αναφέρθηκε το πρόβλημα την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο, αλλά εν τω μεταξύ έγινε συζήτηση στον προπολογισμό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπως γνωρίζετε, και θα ήθελα να ξέρω αν έχετε προχωρήσει τον προβληματισμό σας κυρίως όσον αφορά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνομικής Δυνάμης που είναι ε, αφορά άμεσα την ασφάλεια των πολιτών που είναι προτεραιότητα και θεμελιώδης δικαίωμα. Θα ήθελα λοιπόν να μοιραστείτε μαζί μας, αν δεν τα παρουσιάσατε και στο συγγνώμη, αν δεν το άκουσα, αν δεν το αναφέρατε λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι σκέψεις σας όσον αφορά ε, τη διατήρηση ΕΠΟΛ και τη δημιουργία της αστυνομίας ε, και για τον προπολογισμό του Ευρωπόλ και ε, η δημιουργία του κέντρου καταπολέμησης του εγκλήματος του κυβερνοχώρο που θα δημιουργηθεί τον Ιανουάριο. Για τον προπολογισμό λοιπόν του Ευρωπόλ και του Eurosys. Αν μπορείτε να μου δείτε τα σε αυτά. Ευχαριστώ. Πριν επιστρέψουμε στην Επίτροπο, που σίγουρα σημείωσε δεόντως όλες τις ερωτήσεις που ετέθησαν, ίσως το Συμβούλιο επιθυμεί να πάρει το λόγο. Ίσως επειδή άργησα μίλησε το Συμβούλιο. Όχι. Θέλετε να μιλήσετε, δεν είστε υποχρεωμένοι. Αν δεν θέλετε. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Επίτροπος παρουσίασε την βασική πρόοδο που έγινε. Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν πολλά για να προσθέσουμε. Υπό αυτή την έννοια επιστρέφω το λόγο στην Επίτροπο. Σας ευχαριστώ. Έχετε το λόγο, κύριε Επίτροπε. Thank you very much for your question. Σας ευχαριστώ θερμά για τις ερωτήσεις και για τα σχόλιά σας. Θα προσπαθήσω να δώσω όσο πιο ακριβείς απαντήσεις γίνεται. Καλά. Αν το μικρόφωνο αυτό καλύτερο, να το χρησιμοποιήσω. Σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματο Στοκχόλμη, κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα υποβάλει μια ειδική έκθεση για το θέμα αυτό. Γιατί είχαμε πολλέ εκθέσει αξιολόγηση ήδη. Την ετήσια έκθεση για την μετανάστευση και το άσυλο, για την εσωτερική, στρατηγική εσωτερική ασφάλεια, για το Σέγγεν, για την πάταξη τη διαφθορά και ούτω καθεξής. Δεν θέλουμε επικάλυψη λοιπόν των προσπαθειών και των εκθέσεων αυτών. Ε, θα δοθούν για τις εσωτερικές υποθέσεις ε, ίσως κατάλογοι, ένας κατάλογος ε, για την πρόθεση των εργασιών. Σε ό,τι αφορά το Europol, γιατί πολλοί μίλησαν για το καταστατικό της Europol. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, θα υποβληθεί στις αρχές του νέου έτους, όπως είχαμε υποσχεθεί. Θέλουμε να ενισχύσουμε την προστασία των δεδομένων, να αυξήσουμε την δημοκρατική λογοδοσία η μικρή καθυστέρηση οφείλεται στις ε, δημοσιονομικές περικοπές και τους περιορισμούς και μετά την αποτυχία του προηγούμενου Σαββατοκύριακου θα είναι ακόμη πιο ε, δεινή η κατάσταση και η δημοσιονομική πίεση. Θέλουμε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα και με περικοπή 5% δύσκολο το βλέπω. Γι' αυτό προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικού τρόπου να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα του προγράμματο. σω συγχωνεύσουμε το διοικητικό προσωπικό με τη Europol. Κάνουμε κάποιου ε, υπολογισμού και με τη ΣΕΠΟΛ και με το Συμβούλιο και ανάλογα και με την έκβαση των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό θα υποβάλουμε σχετική πρόταση. Πάντως εμείς θέλουμε μια, ένα ισχυρό σύστημα ε, εκπαίδευσης ε, των αστυνομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τους πόρους για να χρηματοδοτήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα κατάρτισης. Καθυστερήσεις για το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν το 2. Κύριε Κουέλιο, εγώ δεν έχω Πληροφορίε η στοιχεια για άλλε χώρε Εμείς οπω η φιλανδια Εμεί εχουμε υλοποιησει το έργο μα με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σα ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη Φιλανδία. Πήγα όχι εγώ προσωπικά, αλλά συνεργάτε μου πήγα στη Φιλανδία πριν από μία εβδομάδα δέκα μέρε, ε, για να γίνει μια αξιολόγηση τη κατάσταση και να δούμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε τι φιλανδικέ αρχέ για να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση που είναι αναπόφευκτη δεν ξέρουμε ποια θα είναι η διάρκεια της, ένα, δύο μήνες παραπάνω, δεν ξέρουμε ποιε θα είναι οι επιπτώσεις αυτής της ε, καθυστέρησης. Πάντως συνεργαζόμαστε και με εμπειρογνώμονες της Φιλανδίας και την επόμενη εβδομάδα θα υποβάλουμε λεπτομεριακή έκθεση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Θα συζητηθεί 5 και 6 Δεκεμβρίου. Θα λάβετε λοιπόν αυτή την ε, έκθεση και φαντάζομαι θα αποσαφινιστεί η κατάσταση ε, που μας θλίβει ιδιαίτερα και λυπούμαστε που φτάσαμε μέχρι εδώ, αλλά δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά το Σέγγεν, σε λίγο θα έρθει ο κύριος Μαντσεβίτσι μετά το Συμβούλιο ε, για να σας ε, ε, ενημερώσει και τις τελευταίες εξελίξεις. Υπάρχει κάποια πρόοδος και γνωρίζετε τη θέση και την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας την παρουσιάσαμε πριν από καιρό δυστυχώς ε, έχει απορριφθεί σε πολλά σημεία. Πάντως ε, και η Κυπριακή Προεδρία κάνει προσπάθειες. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και είναι σημαντικό η κατάσταση να μην παραμείνει αμετάβλητη. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε το Σέγγεν, να εξασφαλίσουμε λογοδοσία, να γίνει πιο αποτελεσματικό και να αποσαφινιστούν οι κανόνες. Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν λειτουργούν όπως θέλουμε τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά το κλείσιμο των συνόρων, που γίνεται σε έκτακτη περίπτωση. Αυτό που προέκυψε από τις πρωινές συζητήσεις, όπως άκουσα τουλάχιστον, είναι ότι ίσως το Συμβούλιο καταλήξει συμφωνία για μία σύσταση ε, της Επιτροπής. Και νομίζω ότι έχει νόημα να συνεχίσουμε αυτές τις ε, συζητήσεις γιατί έχουν ε, αξία, προστιθέμενη αξία. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη στη συμφωνία, πάντως ε, αργά αλλά σταθερά συμβιώνουμε πρόοδο και προσβλέπω σε τέτοια συμφωνία και θα ρίνω τον κύριο Κοέλιο και τους και ηγητές και την κυρία Βέμπερ να συνεχίσουν τις επικοδομητικές τους προσπάθειες για να καταλήξουμε σε λύση. Αυτό περιμένουν οι συμπολίτες μας από εμάς και θα είναι κρίμα να τους απογοητεύσουμε. Σε ό,τι αφορά την πλήρη ένταξη στο Σέγγεν της Ουρμανίας και Βουλγαρίας, ναι κυρία Αντσίου, το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τεχνική άποψη είναι έτοιμες οι χώρες να ενταχθούν πλήρως. Είμαστε υπέρ της ε, λύσης σε δύο φάσεις. Δυστυχώς ε, η απόφαση του Συμβουλίου ήταν διαφορετική και ε, δεν έχει οριμάσει ακόμη το θέμα. Σε ό,τι αφορά το πακέτο για τα έξυπνα σύνορα, Smart Borders, θα υποβληθεί ο Σονούπο, έχετε και το παρέλειψα, αλλά αποτελεί σημαντικό τμήμα της προσπάθειάς μας να εξασφαλίσουμε πιο εύρυθμη λειτουργία των σύνορων, να διευκολύνουμε είσοδο ε, των ε, προσώπων που θέλουν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ελέγξουμε όσου προσπαθούν ε, παράνομα να εισέλθουν. Τώρα, για τα κονδύλια. Όπως και με πολλά άλλα θέματα, το ρώτησε και ο κύριος Παπα-Νικολάου για το Frontex και για την ΕΑΣΟ. Είχαμε προτείνει αύξηση του προπολογισμού και για την ΕΑΣΟ και για το Frontex, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα, θα, θα καταλήξουν οι συζητήσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γι' αυτό και δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω σήμερα. Κύρια Βέμπερ και κυρία Γκυγιόμ, ρωτήσατε τι γίνεται με τη λαλληλεγγύη. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι δυστυχώς σπανίζει αυτή τη στιγμή η αλληλεγγύη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σίγουρα δεν είναι το πρώτο, η πρώτη μας προτεραιότητα, γιατί τα κράτη-μέλη ασχολούνται με άλλα θέματα. Βέβαια είναι η σημαντικότερη κρίση που είχαμε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί άνθρωποι δεινοπαθούν, εντείνεται ο κοινωνικός αποκλεισμός σε πολλά κράτη-μέλη και μάλιστα υπάρχει μια έξαρση της ξενοφοβίας και του λαϊκισμού. Και αυτό συζητάται μερικέ φορέ στο Συμβούλιο. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι και πιο θετικοί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρά την κρίση είμαστε, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για ένα σύστημα ασύλου που θα είναι καλύτερο από το σημερινό, θα ενισχύσει τις προδιαγραφές, θα εξασφαλίσει καλύτερη προστασία και θα, μπορέσει, θα επιτρέψει στις χώρες να λάβουν τις ευθύνες τους για όσους θέλουν να εισέλθουν και όσους ζητούν ε, προστασία στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλησιάζουμε σε συμφωνία και ήταν πολύ χρήσιμες οι εργασίες αυτές. Και σε μεγάλο βαθμό χάρη στη Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην προσπάθεια χώρων μελών συνεχίζουμε την πρόοδο. Είναι δύσκολη η της ελεγγύης αυτή τη στιγμή. Έχει δειχθεί μεγάλη ελεγγύη προς την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και οικονομικά και στο συγκεκριμένο τομέα και Κυρία Βέμπερ, θα συναντηθώ με τον κύριο Μιλντερ για να ενημερωθώ για την αποστολή αυτή. Νομίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη λίγο ή πολύ συμβάλλουν στην υποστήριξη της Ελλάδας με χρήματα, με εμπειρογνώμονες, με τεχνογνωσία. Ε, όλοι, όλοι οι οργανισμοί έχουν δώσει το παρό στην Ελλάδα για να βοηθήσουν. Έχουμε και ε, διεθνείς οργανισμούς και την υπατερμοστία του ΟΗΕ ε, και καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για να βοηθηθεί η Ελλάδα και φυσικά έχουμε ακόμη πολύ έργο να πραγματοποιήσουμε και μερικά κέντρα κράτησης ε, θα κλείσουν αργότερα. Θα το επισημάνω αυτό στον ε, Υπουργό που θα συναντήσω σε λίγες μέρες. Πάντως υπάρχει πρόοδος και η κυβέρνηση εξετάζει έναν θεωρημένο σχέδιο δράση σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σαφεί ποσοτικοποιημένου στόχου που θα αξιολογούνται τακτικά. Και το θέμα αυτό επανέρχεται τακτικά στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Εξετάζουμε την πρόοδο ή την έλλειψη πρόοδου στην Ελλάδα. Υπάρχει πρόοδο ότι αφορά την πρόσληψη προσωπικού, τη σταθερή ε, δημιουργία ενό ε, συστήματο ασύλου που θα εξασφαλιστεί πρόσβαση στους ετούντες. Φυσικά από άποψη εξασφάλιση των συνθηκών πολλά πράγματα θα γίνουν ακόμη και υπάρχει και το πρόβλημα της ε, βιοπραγιέ κατά των μεταναστών. Αυτό είναι οξύ πρόβλημα. Αλλά σίγουρα όσο εντείνει και η Ελλάδα τις προσπάθειές της, τόσο θα ενισχύεται και η αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Και το θέμα της απορρόφησης. Ε, υπάρχει βελτίωση, υπάρχει καλύτερο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων Υπουργείων και Τμήματων στην Ελλάδα, ώστε να δημιουργηθεί μια καλύτερη εντύπωση για το πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τι ανάγκε. Θα υπάρξουν κονδύλια για την Ελλάδα και τώρα και στο μελλοντικό προπολογισμό. Δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό λοιπόν, είναι θέμα και με τι συνθήκε κράτηση σε μερικά κέντρα. Πάντω θα συνεχιστούν οι προσπάθειε για αρκετό καιρό και η συνεργασία με την Ελλάδα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Τώρα, η αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά ένα υποχρεωτικό σύστημα μετεγκατάσταση δεν υπάρχει καμία απολύτως προοπτική και πιθανότητα να συμφωνήσει το Συμβούλιο σε κάτι τέτοιο. Μόνο δύο χώρες είναι υπέρ. Και στο Λουξεμβούργο, σε ένα γεύμα εργασία, συζητήσαμε το θέμα τη αξιολόγηση του Γιουρίμα. Θα αντιλήσουμε κάποια συμπεράσματα, θα διδαχθούμε από τα παθήματά μα. Θα δούμε πώς θα βελτιώσουμε το σύστημα. Θα συνεργαστούμε φυσικά και με τις Μαλτέζικες Αρχές για τη διαδικασία επιλογής και το καθεξής. Θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια μαθήματα και υποβάλαμε την πρόταση για ένα προαιρετικό σύστημα, γιατί δεν υπάρχει καμία υποστήριξη για ένα υποχρεωτικό σύστημα. Πάντω, έστω και με θελοντικό σύστημα, θα δημιουργήσουμε κάποια ενάψματα στα κράτη-μέλη, θα ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη και με οικονομικά κίνητρα για να εφαρμόσουν το σύστημα. Και μια κλίδα κατανομή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει υποστήριξη ούτε για κλίδα κατανομή στο Συμβούλιο. Και ευελπιστούμε ότι θα επανέλθει κάποια στιγμή η αλληλεγγύη όταν αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο φως στην άκρη του τούνελ σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση. Πρόεδρε, προσπαθώ να διαβάσω τις σημειώσεις μου. Κυρία Γκυγιόμ, συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχουν κάποια στοιχεία στο πρόγραμμα Στοκχόλμης, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Μας μένει περίπου 1,5 χρόνος μέχρι τις ευρωεκλογές. Έχουμε κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας το πρόγραμμα Στοκόλμης συνετάχθη σε άλλες εποχές, άλλο πνεύμα, όπου ξεκινούσε η κρίση, αλλά δεν έχει τις διαστάσεις που έχει τώρα. Υπήρχε δυνατότητα να συντάσει κανείς προτάσεις σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης αλληλεγγύης. Όσον αφορά την ένταξη, όπως αναφέρατε, κάνουμε αρκετά πράγματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν την αρμοδιότητα να θεσπίσουν νομοθεσία, αλλά τακτικά ε, δημιουργούνται διάφορα φόρα όπου διάφοροι ντόπιοι φορεί συναντώνται, ανταλλάσσουν απόψεις, συστάσεις. Έχουμε το εγχειρίδιο, το handbook, έχουμε στο σελίδα και συζητούμε το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό. Συμφωνώ μαζί σας, πράγματι πρέπει να γίνουν περισσότερα όσον αφορά τα δικαιώματα των μεταναστών Εκεί θα είμαι ανοιχτή προς συζήτηση. Πώς μπορεί να επιτευχθεί πρόοδο. Είναι κάτι μελλοντικό. Πώς να αντιμετωπίσουμε τα δικαιώματα των μεταναστών ολιστικά για όλους. Καλή ιδέα για το μέλλον. Δεν κάναμε αρκετά πράγματα. Για την ώρα, όπως είπαν και οι συνάδελφοί σα πρέπει να εστιαστούμε στην ολοκλήρωση του πακέτου του ασύλου, να επαγρυπνούμε για την εφαρμογή πριν κάνουμε και άλλες προτάσεις. Αλλά ας κάνουμε και μία χάρτα δικαιωμάτων των μεταναστών. Είναι κάτι προς την, που πρέπει να το εξετάσουμε ερωτικά μετά τη Στοκχόλμη. Κυρία Ματιού, σας είπα αυτά που ξέρω για την ώρα όσον αφορά τη ΕΠΟΛ. Κυρία Ιντβέλτ για τον Καναδά, ναι και εμείς έχουμε απογοητευτεί για την έλλειψη πρόοδου, ξέρουμε τις ανησυχίες που εκφράσατε. Όλοι εκφράσατε στην τελευταία συνεδρίαση με τον κύριο Πρίμπε που παρουσίασε την κατάσταση, συμφωνώ με τι περισσότερε ανησυχίε, τι διαβίβασα στου Καναδού. Ελπίζουμε να έχουμε νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Χρειάστηκε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι άκρο απογοητευτικό. Και ελπίζω πολύ σύντομα να προχωρήσουμε για να υπάρξει νομική σαφήνεια όσον αφορά την διατήρηση των στοιχείων. Το συζητήσαμε στην Ολομέλεια πριν από λίγο. Δεν συνέβησαν πολλά έκτοτε, εκτός από κάτι που σας υποσχέθηκα και δεν πραγματοποιήθηκε ακόμα. Πληροφορίες που μας στέλνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τη χρήση αυτού. Λάβαμε περισσότερες πληροφορίες και όταν συζητώ με μέλη, όλοι εκτός από ένα-δύο δεσμεύονται ε, να συμμορφωθούν την οδηγία για την διατήρηση των στοιχείων και αν λένε κάτι άλλο σε εθνικό επίπεδο, είναι πολύ παράξενο τη δηλαδή, συνεδρία του Συμβουλίου. Όλοι υποστηρίζουν ένθερμα την οδηγία και θέλουν να την επεκτείνουν μάλιστα και όχι να, την να απαλλαγούν από αυτή. Κύριε Έντβελτ, δεν λέω ότι η Ολλανδία δεν συμφωνεί, αλλά ότι είναι ανεπαρκή σε εφαρμογή. Η αστυνομία χρησιμοποιεί τα στοιχεία χωρίς να τηρεί τους κανόνες. Ε, πράγματι, λέει κύριε Επίτροπος, η άνηση αυτή και διαφορετική ερμηνεία και εφαρμογή της οδηγίας για τη διατήρηση των στοιχείων είναι κάτι που ενετόπισε και επέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό χρειάζεται αναθεώρηση. Όμω πρέπει να γίνει αυτό ταυτόχρονα με την ε, αναθεώρηση <laughs> Την οδηγία για την προστασία των ηλεκτρονικών στοιχείων, προστασία της ιδιωτικής ζωής. Υπάρχει ένα κενό εκεί, γιατί λέει ότι μπορεί, η νομοθεσία μπορεί να συλλέγονται ε, στοιχεία για άλλους σκοπούς. Για την πρόταση TFTS, αρχές του επόμενου έτους θα επιστρέψουμε, θα σας δώσουμε πληρέστερη παρουσίαση των διαφόρων υπαρχουσών εναλλακτικών. Ο κ. Πρεβό και ο κ. Μασχοβής ήταν εδώ πριν από λίγο καιρό να σε εξηγήσουν για τα τα στοιχεία, όπως είπα στην εισαγωγή μου, τα API μάλλον, είναι πιο περίπλοκο το θέμα. Υπάρχουν πολλές επικαλύψεις νόμων σε εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να δούμε ποια λύση μπορούμε να βρούμε. Και υπόσχομαι να επανέλθω συντομότατα με πιο συγκεκριμένη ιδέα. Πράγματι κάτι πρέπει να γίνει. Το ερώτημα είναι τι, αλλά και πώς. Εμπλέκονται πάρα πολλές χώρες. Σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να υπάρξουν συμφωνίες. Όλα αυτά πρέπει να εξεταστούν νομικώς. Διαφάνεια. Σημαντική πράγματι. Ενθαρρύνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν γέννη να διαδραματίσει το ρόλο του, να ελέγχει, να παρακολουθεί. Αναφερθήκατε συγκεκριμένα στο TFTP, τη συμφωνία SWIFT. Η διαφάνεια δεν μπορεί να εφαρμοστεί ομοιόμορφα γιατί μιλάμε για απόρριτες πληροφορίες. Άρα χρειάζεται συγκεκριμένη προσέγγιση. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις μαζί με τους Αμερικανούς ομολόγους μας. Εκάλυψα όλα τα ερωτήματα, θα ρω, Πρόεδρε. όχι από τα κρατημέλη, από τα μέλη τη Επιτροπή ε, ε, Πολιτικών Ελευθεριών, λέει ο Πρόεδρος. Συγγνώμη, λέει η κυρία το ξέρω, το ξέρω. Ζητώ συγγνώμη. Η περασμένη εβδομάδα ήταν πολύ δύσκολη. Μέλη λοιπόν, τα μέλη της Επιτροπής ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Ευχαριστώ πολύ που, για τις προσπάθειές σας να θέματα που ετέθησαν σύμφωνα με το πώς γνωρίζετε τα θέματα και μάλιστα απαντήσατε και ε, μέσα στο χρονικό περιθώριο που είχαμε προβλέψει, μια μισή ώρα δηλαδή, για την απογευματι... στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Ε, υπάρχει κάποιο μέλος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που θέλει να επανέλθει, να κάνει και νέα ε, εξέταση της Επιτρόπου. Αν όχι, θα σας ευχαριστήσουμε, Επίτροπε Μάλμστρομ. Ε, όπως πάντα που έρχεστε εδώ πρόθυμοι να μοιραστείτε μαζί μας τις λεπτομέρειες των ε, προγραμμάτων που έχουν τεθεί για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Και τώρα, ε, στις 18, πρέπει να ανακοινώσω ότι στις 18 Δεκεμβρίου θα έρθει η Αντιπρόεδρος Ραντίν για να συζητήσει μαζί μας το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και την ενδιάμεση αξιολόγησή του, η επανεξέτασή του στον τομέα της δικαιοσύνης όπως κάναμε και στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ και τώρα πάω να εξετάσω την ε, ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. I am announcing that Το επόμενο θέμα, παρακαλώ να κάνω μια ανακοίνωση. Δεν έχω σφυράκι. Θέλω την προσοχή σας όμως. Το επόμενο θέμα είναι του κυρίου Μανσερβισή που θα παρουσιάσει ε, τις εσωτερικές υποθέσεις. θα γίνει μετά από το πεντάλεπτο διάλειμμα γιατί δυσκολεύεται να μπει στο κτίριο του Κοινοβουλίου λόγω του αποκλεισμού στην ε, περικείμενη περιοχή από τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για την ε, κατάσταση της ε, αγροτικής γεωργικής πολιτικής. Πέντε λεπτά διάλειμμα. Καλησπέρα σας κύριε Μασερβίση. Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε και πάλι στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Μόλις ολοκληρώσαμε την ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Μάνστρομ, είστε έτοιμος να περάσουμε αυτή αμέσως στο επόμενο σημείο. Που αφορά ένα θέμα ιδιαίτερα προσφυλές και σε και τη Γενική Διεύθυνσή σας δηλαδή τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για τον έλεγχο της εφαρμογής του κεκτημένου Σέγγεν. Η συγγετής μας για το θέμα αυτό είναι ο κύριος Κάρλος Κοέλιο. Ένα θέμα που φυσικά είναι συναφέ και με το σημείο 5, τροποποίηση του κανονισμού 562 του 2006, με σκοπό τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε έκτακτες περιπτώσεις. Έχουμε εισηγήτρια για το θέμα αυτό την κυρία Βέμπερ. Είναι αλληλένδετα τα δύο θέματα και φυσικά άπτονται του πακέτου διακυβέρνηση του Σέγγεν. Το θέμα αυτό θα το εξετάσουμε διεξοδικά μετά το Συμβούλιο ε, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ιουνίου που αποφάσισε να τροποποιήσει τη νομική βάση από το άρθρο 70 δημιουργώντας ε, μία θεσμική αντιδικία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα με την δική μας Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών. Η διάσκεψη Προέδρων μας ε, ε, σύστησε να ξεκινήσουμε διερευνητικές επαφές με την Κυπριακή Προεδρία προκειμένου να καταλήξουμε σε κοινέ θέσει για το θέμα αυτό και οι δύο συγκητές μας, Κοέλιο και Βέμπερ, είχαν πολλαπλές επαφές με την Κυπριακή Προεδρία, με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τους και συγκητές. και θα δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα. Θα έλεγα λοιπόν να δώσουμε πρώτα το λόγο στους συγκητές μας, Κοέλιο και Βέμπερ. Μετά θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μασερβίση, και κατόπιν την Κυπριακή Προεδρία. Κύριε Κοέλιο, έχετε το λόγο πρώτα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς, είχαμε πολύ άριθμες συναντήσεις προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποια κοινά σημεία και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αρκετέ αδρέ γραμμές. Καταρχήν, συμφωνούμε ότι Σέγγεν σημαίνει ευρωπαϊκή προσέγγιση, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να σεβαστούμε την εθνική κυριαρχία. Γιατί υπάρχουν πολλές εξουσίες και αρμοδιότητες ε, ε, που αφορούν τα τον έλεγχο των συνόρων και είναι αποκλειστικά εθνικές αρμοδιότητες. Στην πράξη όμως, όταν μιλούμε για το Σέγγεν, ε, εννοούμε τα κοινοτικά σύνορα, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε επίσης συμφωνία ως προς το γεγονός ότι χρειαζόμαστε έναν κοινοτικό μηχανισμό, έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό και στην ε, διαδικασία αξιολόγηση πρωτοστατεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στενή όμω ανάμειξη και των κρατών μελών. Δηλαδή, οι ομάδε των εμπειρογνωμών θα έχουν επικεφαλή σε έναν εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φυσικά οι εμπειρογνώμονε είναι εμπειρογνώμονε των κρατών μελών και η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη για να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη που είναι εκ των όνων κάνει προϋπόθεση για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του Σέγγεν. Πιστεύω ότι και Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούν ως προς, τον, ως προς την ανάγκη να δοθεί επαρκής ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Συμβούλιο. Γιατί διαπιστώσαμε ότι η διατύπωση που θέτησε το Συμβούλιο δεν ήταν αυτή που είχαμε ζητήσει εμείς. Αλλά παρόλα αυτά δεν πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα γιατί η Κυπριακή πρωτοβουλία, η Κυπριακή Προεδρία μας δήλωσε πολλαπλώς ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε ειδικού κανόνες για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες, για τις απόρριτες πληροφορίες, με ειδικού κανόνες για την πρόσβαση σε αυτές. Όπως ξέρετε, το μείζον πρόβλημα ήταν το νομικό πρόβλημα, γιατί το Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιεί τη νομική βάση από το άρθρο 77 στο άρθρο 70. Μετά από εκτενείς συζητήσεις και μετά την πρόταση και τη γνωμοδότηση της νομικής μας υπηρεσίας, συμφωνούμε τελικά με την ιδέα της θέσπης μιας ρήτρας γεφύρωσης, δηλαδή μιας ρήτρας στον κώδικα συνόρων ε, του Σέγγεν που θα ε, κάνει τη σύνδεση με το μηχανισμό αξιολόγηση του Σέγγεν για να μην χρειαστεί να αλλάζει κάθε φορά ε, το, ο κώδικας του σύνορου του Σέγγεν για, το οποίο, για τον οποίο ισχύει συναπόφαση. Η νομική αυτή λύση εξετάστηκε και από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Α με διορθώσει η Ρενάτε Βέμπερ αν κάνω λάθο. Πάντω, εγώ αποκόμισα από την τελευταίο τριμερή διάλογο την εντύπωση ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Αλλά όταν μιλούμε για το bridging clause, τη ρήτρα γεφύρωση, εννοούμε ουσιαστικά την ενίσχυση τη διατύπωση. Και ο ακριβή τρόπο. Ε, η ακριβή διατύπωση για αυτή τη ρήτρα γεφύρωσης είναι να διασκεδαστούν ε, οι ανησυχίες μας και να ληφθούν υπόψη τα σχόλιά μας. Πριν από λίγο ε, εξετάσαμε με την Επίτροπο Μάρμουσον το θέμα της ε, απόφασης για τη σύσταση. Το Συμβούλιο έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κάποιε αλλαγέ στη διακυβέρνηση του Σέγγεν προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια και να προβλεφθεί μία νέα ρήτρα για την επανειφορά των ελέγχων στα σύνορα. Το Κοινοβούλιο είπε από την αρχή ότι δεν θέλουμε να παρακολύσουμε την ελεύθερη διακίνηση, αλλά θα μπορούσαμε να δεχτούμε την ε, εισαγωγή μια ρήτας επαναφοράς ε, των ελέγχων ω συνέπεια του μηχανισμού αξιολόγησης. Τελικά, τελευταία στιγμή, το Συμβούλιο υπέβαλε μια άλλη ιδέα όχι μια απόφαση, ε, όχι απόφαση για την επαναφορά των, σύνορα, ελέγχων στα σύνορα, αλλά μια σύσταση μόνο. Δηλαδή, αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν σοβαρά ε, προβλήματα με τον έλεγχο των σύνορων σε ένα κράτος ακόμη και αν το σύνολο της, ε, του χώρου Σέγγεν αποφασίσει, όλες οι χώρες του Σέγγεν αποφασίζουν ότι δεν είναι αξιόπιστη αυτή η έλεγχη στο συγκεκριμένο κράτος και υπάρχει ανάγκη επαναφορά των ε, ελέγχου στα σύνορα. Παρ' όλα αυτά, οι χώρε δεν μπορούν να λάβουν απόφαση και να υποχρεώσουν επαναφορά των σύνορων, αλλά μόνο σύσταση μπορούν να υποβάλουν και να και στι χώρε να δεχτούν ή όχι αυτή τη σύσταση στι ενδιαφερόμενε. Εγώ έδωσα το παράδειγμα τη πατρίδα μου τη Πορτογαλία. Είπα, φανταστείτε ότι η Πορτογαλία έχει ένα πρόβλημα. Ότι η Πορτογαλία δηλαδή δεν μπορεί να λύσει μόνη της το πρόβλημα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ό, τα υπόλοιπα κράτη διαπιστώνουν ότι η Πορτογαλία έχει πρόβλημα με τον έλεγχο στα σύνορα και αποφασίζουν να επαναφέρουν τους ε, ελέγχους. Αν δεν έχουμε να κάνουμε με απόφαση αλλά με απλή σύσταση, τι θα συμβεί. Μερικές χώρες θα δεχτούν τη σύσταση και θα επαναφέρουν τους ελέγχους, ενώ άλλες δεν θα τη δεχτούν. Αν όμω θέλουμε να είναι ασφαλής ε, η ζώνη Σέγγεν, ο χώρο Σέγγεν, δεν θα έχουμε αποτελεσματικότητα στο σύστημα αν μόνο μερικές χώρες δεχτούν τη σύσταση και άλλες όχι. Γιατί είναι προφανές ότι οι άνθρωποι θα περνάνε από τις ε, χώρες που δεν έχουν επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορα, που είναι ανοιχτά τα σύνορα. Άρα παρακάμπτουμε το σύστημα Σέγγεν. Τελικά, είπαμε να δεχτούμε από την Κυπριακή Προεδρία μια γραπτή δήλωση γιατί μετά από όλους αυτούς τους ε, διαλόγους και τους τριμερείς διαλόγους ε, να υποβληθεί πρόταση με τη συγκεκριμένη διατύπωση που μπορεί να δεχτεί το Κοινοβούλιο και, με και τις διατυπώσεις που δεν μας βρίσκουν σύμφωνους ε, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σαφή αξιολόγηση. Πάντως τα βασικά προβλήματα, τα βασικά προσκόμματα είναι αυτά που σας ανέλησα. Ευχαριστώ. Κυρία Βέμπερ, η σειρά σας τώρα. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μανσερβίση που ήρθατε να μας δείτε στην Επιτροπή μας. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Κοέλιο. Να υπογραμμίσω ένα πράγμα μόνο και θα το λέω ξανά και ξανά αν χρειαστεί. Όταν άρχισε η όλη υπόθεση, η βασική ιδέα ήταν να βελτιώσουμε τον υφιστάμενο μηχανισμό. Αλλιώς δεν θα είχε υποβάλει καινούρια πρόταση κομισιόν αν δεν το είχε αυτό υπόψη της. Και το Κοινοβούλιο προφανώς ήθελε μια ένα τέτοιο επίτευγμα σημαντικό όπως ο χώρος του Σέγγεν να διοικείται και να ε, διέπεται από κοινοτική προσέγγιση γιατί είναι ολονών και όχι των μεμονωμένων κρατών μελών. Από την άλλη πλευρά είναι αλήθεια ότι ενίοτε είναι δύσκολο να δικαιολογήσουμε την αλλαγή ενός συστήματος αν η αξιολόγηση είναι ότι το σύστημα πήγε καλά, που αυτή ήταν η αξιολόγηση της Κομισιόν. Όχι μόνο δεν άρχισαν ποτέ διαδικασίες επί παραβάση, αλλά οι αξιολογήσεις ε, ήταν θετικές. Καταλαβαίνω λοιπόν και την αντίσταση από τα κράτη-μέλη που λένε ότι δεν θέλουμε τέτοια δραματική αλλαγή για ένα σύστημα το οποίο τα πήγε πολύ καλά. Αυτή όμως είναι η θέση του Συμβουλίου. Η θέση του Κοινοβουλίου ήταν να εγκρίνουμε την πρόταση της Κομισιόν και ειλικρινά νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι κάναμε δεκάδες άτυπες ε, ανεπίσημες συναντήσεις, επίσημους τριμερείς ε, διαλόγους και συζητήσαμε μέχρι και το τελευταίο κόμμα των προτάσεων αυτών. Και τώρα αντιλαμβανόμεθα ότι είμαστε αντιμέτωποι σε μια κατάσταση που μας κάνει να πιστεύουμε ότι όλη αυτή η δουλειά των τελευταίων μηνών λίγος πολύ απέβει μάταια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το σύστημα δεν είναι ότι βελτιώνεται με μεγαλύτερη ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που βεβαίως είναι ευπρόσδεκτη, αλλά το σύστημα θα βελτιωθεί μέσα από αποφάσεις όταν αυτό δεν λειτουργεί, όταν υπάρχει πρόβλημα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, έχουμε κολλήσει στις δύο διαφορετικές θέσεις. Εμείς θέλουμε να ληφθεί απόφαση και το Συμβούλιο λέει όχι, δεν πρόκειται για τη λήψη απόφασης ούτε από το Συμβούλιο ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ληφθεί και από το Συμβούλιο η απόφαση. Είμαστε πρόθυμοι να υποχωρήσουμε ε, από την κοινοτική προσέγγιση που θα πρόβλεπε την Κομισιόν. Αλλά από ό,τι καταλάβαμε από το τελευταίο τριμερή διάλογο, δεν πρόκειται γι' αυτό. Δεν είναι δηλαδή ούτε απόφαση. Πρόκειται για σύσταση, λένε τώρα. Και όχι από τα ε, υπεύθυνα κράτη-μέλη, αλλά από τα άλλα κράτη-μέλη, τα υπόλοιπα. Βεβαίως, περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τι προτάθηκε σήμερα που θα μας το πει ο κύριος Μανσερβίση. Δεν θέλω να πω αυτή τη στιγμή ότι εμείς είμαστε άκαμπτοι στην προσέγγιση μας, αλλά πρέπει να πούμε δύο πράγματα για να είμαστε εντάξει. Πρώτον, οι δύο εκθέσεις θα πρέπει να θεωρηθούν πακέτο με την έννοια ότι οι διαπραγματεύσεις επί της μιας έκθεσης θα πρέπει να έχει κάποια συν και για την άλλη έκθεση. Επίσης, ε, πρέπει να πούμε ότι είμαστε ανοιχτοί και πρόθυμοι να συνεχίσουμε τη συζήτηση και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στο βαθμό που έχουμε την αίσθηση ότι αυτό που θα ψηφίσουμε θα αποτελεί γνήσια βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Αλλιώς, α, ειλικρινά αναρωτιέμαι αν έχει νόημα να μπούμε σε όλον αυτό τον κόπο. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κυρίος Μανσερβίση και η Κυπριακή Προεδρία θα, μας, θα λάβουν το λόγο πριν δώσουμε το λόγο στα υπόλοιπα μέλη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Ακούω. Προσπαθώ να ακούσω τι απόψεις που επικρατούν και να δω αν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στα εφιστάμενα και στο τι μπορούμε να έχουμε στο μέλλον. μπείτε στην κατάσταση που κρατούσε πέρσι, που είναι ίδια με τη φετινή. Υπάρχει ένα πρόβλημα που προέρχεται και από το εξωτερικό και από την αδυναμία ενός κράτους μέλους να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν το Σέγγεν. Και για να καλυφθεί το κενό υπάρχει μία διαδικασία τα που την εφαρμόζουν οι υπάλληλοι και ακολουθούν διαδικασία που ενεκρίθη σε σημείο Α στο Συμβούλιο χωρί συζήτηση με του ε, διαφόρου ενδιαφερμένου και, το Κοινοβούλιο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρατηρητή. Αυτή η κατάσταση επικρατεί όσον αφορά την ανάλυση για τον εντοπισμό ενδεχομένων προβλημάτων. Και δεύτερον, όσον αφορά την εξωτερική κρίση που μπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους, δεν έχουμε κάποιο κοινό μηχανισμό για λήψη απόφασης. Είδατε, είδαμε, τι συνέβη πέρσι σε κάποια στιγμή. Δεν κρίνω, αλλά δεν ήταν η καλύτερη εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή που προβλήθηκε. Αντιμετωπίζοντας ένα συλλογικό πρόβλημα που, που αντιμετώπισε το Σέγγεν, που είναι κοινό αγαθό, αντιμετωπίστηκε ποικιλοτρόπως από κάθε χώρα ξεχωριστά. Εφαρμόστηκαν εθνικές πολιτικές. Αυτό συμβαίνει αν δεν υπάρχει ένας μηχανισμός για κοινή λήψη απόφασης. Κάθε κράτος αποφασίζει ανάλογα με την κρίση του και τη διάγνωσή του για το πρόβλημα. Άρα κατακαιρματισμένη προσέγγιση που δεν αντικατοπτρίζει τον κοινό χώρο Σέγγεν. Και η προσέγγιση αυτή είναι εντελώς αναποτελεσματική, για, διότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του δικού του κομματιού Σέγγεν. Δεν μιλάμε για εθνικά σύνορα εδώ. Όταν μιλάμε για το Σέγγεν, συζητάμε του τι μέσο διαθέτουμε για να υπερασπιστούμε με αξιόπιστο τρόπο το Σέγγεν. Αξιόπιστο τι εννοώ. Όπως ξέρετε πολύ καλά, θέλουμε οι πολίτες να απολαμβάνουν την ελευθερία, αλλά και να αισθάνονται ότι προστατεύονται από ένα κοινό μηχανισμό, που θα αντιμετωπίζει ενδεχόμενα προβλήματα. Προβλήματα που αφορούν όλο το χώρο Σέγγεν. Αυτό αντιμετωπίσαμε πέρσι και αυτό αντιμετωπίζουμε τώρα. Αν συμβεί ξανά κάτι, ξανά στην ίδια κατάσταση θα βρισκόμαστε. Εξού και οι προτάσεις μας. Η πρότασή μας μάλλον. Ο μηχανισμός από διακυβερνητική συνεργασία με εθνική λήψη απόφασης που προστατεύει μόνο ένα κομμάτι του χώρου, αυτό είχαμε πριν, θέλουμε να το μετατρέψουμε σε ένα κοινοτικό σύστημα. Αυτή την προσέγγιση ακολουθήσαμε. Αντιμετωπίσαμε κάποιο κίνδυνο, αλλά το κάναμε. Κοντολογής καταλήξαμε σε απόφαση στο Συμβούλιο για τα δύο μέσα για την αξιολόγηση Σέγγεν και για τον ε, μεθοριακό κώδικα Σέγγεν. Μετακινήθηκε το κέντρο της βαρύτητας από κοινοτικό μηχανισμό σε ευρυδικό. Κυρίως όσον αφορά το μηχανισμό αξιολόγησης και όσον αφορά την επανεισαγωγή ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα. Άμα δούμε την ουσία όμως, ήδη έγινε ένα βήμα προόδου σημαντικό. Γιατί, γιατί αναγνωρίστηκε σαφώς, αν δείτε την απόφαση του Συμβουλίου, αναγνωρίστηκε λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα από κάθε κράτος. Αναγνωρίστηκε ότι το κοινό μας αγαθό, το Σέγγεν που διαχειριζόμαστε, χρειάζεται μια ανταπόκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο από μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ανεξάρτητα από το μηχανισμό που θα αποφασιζόταν, ακολουθήθηκε διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική ανάλυση. Δεχτήκαμε ότι όταν έχουμε κοινό πρόβλημα χρειαζόμαστε κοινή λύση. Ελήφθη απόφαση τον Ιούνιο. Μετά από αυτό έγινε έξοχη δουλειά από την Κυπριακή Προεδρία. Έπρεπε να χειριστεί απόφαση δανεικής Προεδρίας που επεκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι δεν είχε επιτευχθεί σωστή ισορροπία. Η κυρία Βέμπερ και ο κύριος Κοέλιο έθεσαν το πλαίσιο. Αν πω σε αυτό το πλαίσιο, θα πω ότι ουσιαστικά ακολουθούμε την ίδια προσέγγιση. Αναγνωρίστηκε ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να λάβει χώρα με αυτόν τον τρόπο, τον ελαφρύ του ΣΥΠΗΝ και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει εξολόγηση βάσει στοιχείων. Όλοι έχουν συμφωνήσει από αυτού. Είναι σημαντικό αυτό. Όχι γιατί αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά γιατί είμαστε ένα ανεξάρτητο φορέας, ανεξάρτητος από πλευρά πολιτική. Και για να διατηρήσουμε και επαφή με την τεχνογνωσία την επιτόπια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει ομάδες τον οποίων ηγείται και αναλαμβάνει την ευθύνη, την πολιτική έναντι του Κοινοβουλίου. Αλλά η ομάδα συμπεριλαμβάνει εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη και από φορείς, εμπλεκόμενος. Όπως προανέφερα, ε, έχουμε αποδεχτεί αυτή την προσέγγιση, σημαντικό βήμα πρόοδου. Όλοι κινούμεθα προς την ίδια κατεύθυνση. Όταν εντοπιστούν τα στοιχεία, τι να κάνουμε. Επόμενο βήμα. Προφανώς αυτό ακόμα παραμένει εν μέρει ανοιχτό. Κάποιοι λέγουν ότι υπάρχει σύσταση, άλλοι λέγουν ότι υπάρχει πρόταση με απόφαση του Συμβουλίου. Αν πάμε κατευθείαν στο στόχο, στόχος είναι η δεσμευτική απόφαση. από τη στιγμή που διαπιστώνται τα στοιχεία. Τι χρειάζεται. Όταν ένα θεσμικό όργανο, όπως είναι το Κοινοβούλιο, αποφασίσει περί συστάσεως ή συγκεκριμένης αποφάσεως, κλείνει το ζήτημα. Δύσκολο να αποδείξει κανείς ότι κάτι δεν πρέπει να γίνει. Εδώ συμφωνώ με την κυρία Βέπερ. Είναι ασφαλέστερο όμω να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ληφθεί απόφαση, γιατί είναι πιο ξεκάθαρα πράγματα. Προ τα εκεί πρέπει να κινηθούμε. Όμω μόνο αφού ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα, τι πρέπει να κάνουμε. Και η χώρα έχει το βάρος να απορρίψει μια σύσταση που θα γίνει. Πρόταση για λήψη απόφαση είναι καλύτερη λύση. Το ίδιο και για τον κώδικα των συνόρων Σέγγεν, όπως είπε η κυρία Βέμπερ και ο κύριος Κοέγιο. Τι να πούμε πάνω σε αυτό. Πρώτον, ποιος ο μηχανισμός λήψης απόφασης σε περίπτωση απειλής για το χώρο Σέγγεν και για την εισαγωγή μεθοριακών ελέγχων. Ήδη έχει γίνει το πρώτο βήμα. Αναγνωρίσαμε ότι για να προστατεύσουμε όλη την περιοχή αυτή χρειάζεται συνολική απόφαση. Με μοναμένη απόφαση προστατεύει μόνο ένα κομμάτι Σέγγεν από μια χώρα. Αν υπάρχει πρόβλημα για όλη την περιοχή, χρειάζεται γενική απόφαση. Αυτό αναγνώριση το Συμβούλιο. Σημαντικό. Πώς θα γίνει αυτό. Έτοιμα, σύσταση. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αν υπάρξει πρόβλημα όπως κατά το παρελθόν θα είναι δύσκολο να μην γίνει αυτό που θα έχει συσταθεί. Αν υποβληθεί πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ληφθεί απόφαση, είναι πιο ξεκαθαρά τα πράγματα, γιατί είναι δεσμευτική και σαφή. Uh, uh, uh, λοιπόν, ας πούμε ότι δεν θέλουμε να έχουμε την κατάσταση ότι στην οποία υπάρχει κενό από τη μία και απόφαση από την άλλη. δεν έχουν, μερικά, δεν έχουν περιθώρια ελιγμών τα κράτη-μέλη για τη λήψη απόφαση όταν προκύψει πρόβλημα. Είναι καλύτερο για ασφάλεια δικαίου να έχουμε ένα νομικά δεσμευτικό μέσο που θα χρησιμοποιείται. Το επεξεργαζόμαστε ακόμα. Δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα αυτό, απλώς σκιαγραφώ την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μετά η ρήτρα γεφύρωσης, bridging clause. Είναι μια διέξοδος αυτή. Συνδυάζει την ουσιαστική λύση με το ευαίσθητο νομικό θέμα. Άρθρο 70 που είναι η νομική βάση που αποφάσισε το Συμβούλιο που δεν μας αρέσει και δεν είναι εκεί μας πρόταση. Ταυτόχρονα συνεπάγεται αναγνώριση των προαναφερθέντων. Αν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι υπόλογοι έναντι του Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνουν και συζητούν μαζί με το Κοινοβούλιο τα πορίσματα των αξιολογήσεών μας και αν ο μηχανισμός γεφύρωσης καθορίζει τι θα κάνει ο μηχανισμός αξιολόγησης ώστε να είναι ένα εργαλείο που λειτουργεί σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σέγγεν. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, συνδυάζουμε συμβιβασμό, πολιτικό ρεαλισμό και έτσι η ρήτρα γεφύρωσης αξίζει επεξεργασίας και ανάλυσης για να λάβουμε υπόψη τις διάφορες νομικές συνιστώσεις. Για να επικρατεί μεγαλύτερη σαφήνεια. Έτσι θέλουμε να κινηθούμε για να τα συνδυάσουμε αυτά. Ούτως ώστε η συναπόφαση, η νομική βάση της συναπόφασης να επικρατήσει που είναι και η αφετηρία της χρήσης του μηχανισμού του Σέγγεν. Αν τα καταφέρουμε να κινηθούμε ότι ο τρόπος, πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Με την επιφύλαξη κάποιας μεγάλης πολιτικής αξιολόγησης. Αυτό είναι άλλο θέμα. Διοργανικής φύσεως. Αν καταλήξουμε σε συμφωνία που ανταποκρίνεται σε αυτά που είπε η κυρία Βέπερ, σε ριζική βελτίωση των όσων έχουμε. διότι αυτό είναι το α και το ω, τότε θα είμαστε σε καλή θέση. Εμείς δεν θα συμβιβαστούμε όσον αφορά το δικό μας ρόλο. Αν βάλω τον εαυτό μου στη θέση που βρισκόμασταν πέρσι και χρησιμοποιήσω αυτό το πλαίσιο, βλέπω ότι έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο. Εγώ έτσι βλέπω για την ώρα την όλη κατάσταση. Θα προσπαθήσουμε. ευχαριστώ. Θα προσπαθήσουμε ως συνήθω θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Ας ακούσουμε όμως τον κύριο Κωνσταντινίδη, τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Προεδρίας. Έχετε το λόγο. Και καλό απόγευμα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα εκ μέρους της Προεδρίας αλλά και του Συμβουλίου να εκφράσω τις σερμέμους μου ευχαριστίες προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα προς τους δύο συγγητές των προτάσεων για τη διακυβέρνηση Σέγκεν, τον κύριο Κάρλος Κοέγιο και την κυρία Ρενάτε Βέπερ για την άψογη συνεργασία, ε, καθώς και για την ευελιξία και διάθεση που επέδειξαν για εξέβρεση αποδεχτήσιμη συμβιβαστικής λύσης επί των δύο προτάσεων. Θα ήθελα επίση να εκφράσω τις ευχαριστίες της Προεδρίας προς τον κύριο Μασεβίση για τα καλά του λόγια, αλλά και για την αναγνώριση των επίπονων προσπαθειών που καταβάλλονται από την Προεδρία για επίτευξη σημαντικής προόδου επί των δύο προτάσεων. Θα ήθελα να τονίσω ότι παρόλο που γνωρίζαμε από την αρχή ότι υπάρχουν κόκκινε γραμμέ τόσο από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και από πλευρά Συμβουλίου επί συγκεκριμένων σημείων, εν τούτης είμαι στην ευχάριστη θέση να δηλώσω ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδο και ότι η Προεδρία είναι αισιόδοξη ότι μέσα σε αυτόν το πνεύμα επικοδομητική συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, η επίτευξη συμβιβαστική συμφωνία είναι εφικτή μέχρι τα τέλη τη Κυπριακή Προεδρίας. Να σας ενημερώσω ότι σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Συμβούλιο όπου συζητήθηκαν πιθανές συμβιβαστικές λύσεις ε, στη βάση των διαπραγματεύσεων τριλόγου που πραγματοποιήθηκαν με του δύο εισηγητές. Τα αποτελέσματα τη συζήτηση αυτή στο Συμβούλιο θα αποτελέσουν τη βάση για συνέχιση των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν, ίσως ακόμα και από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Κλείνοντας, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τις ευχαριστίες μου προς τους δύο συγγητές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εντατικές προσπάθειες που καταβάλουν για εξέβρεση συμβιβαστικής συμφωνίας και να σας διαβεβαιώσω ότι η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει με τον ίδιο εντατικό ε, ρυθμό τις προσπάθειες προς το σκοπό αυτό. Σας ευχαριστώ. Now, let's have some floor for discussion. Μάλιστα, κύριε Σεντσίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι οι συνάδελφοι Κάρλο Σκοέλιο και Ρενάτε Βέμπερ μας έκαναν μια πολύ πιστή περιγραφή της κατάστασης. Και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε τεράστιες ε, υποχωρήσεις για να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση. Γιατί θέλουμε ε, μια συμβαστική λύση που θα έχει μια ελάχιστα, μη τι άλλο, ευρωπαϊκή προσθεθέμενη αξία. Αλλά από τις πολυάριθμες αυτές ε, συναντήσεις δεν διαπίστωσα αντίστοιχη προθυμία για πρόοδο και από πλευρά Συμβουλίου. Αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα ατού. Γιατί αν μη τι άλλο είναι ενωμένο, έχει μια ενιαία γνώμη για το θέμα της ε, διακυβέρνησης του χώρου Σέγγεν. Όλες οι πολιτικές ομάδες ε, έχουν την ίδια γνώμη θα πρέπει το Συμβούλιο να αντιληφθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο για διαπραγματεύσει, αλλά έχει και κάποιες κόκκινες γραμμές που δεν μπορεί να τις ξεπεράσει. Για παράδειγμα, ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το μηχανισμό αξιολόγησης είναι σημαντικός. Και το σύστημα κυρώσεων εις βάρος των χωρών που δεν συμμορφώνονται με τον κώδικα των σύνορων Σέγγεν. Επίσης, η επαναφορά των ελέγχων στα σύνορα θα πρέπει να γίνει μετά από διαβούλευση με όλες τις χώρες μέλη. Και φυσικά αυτή η λύση θα πρέπει να είναι η ίστατη λύση. Θα πρέπει επίσης να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική συμφωνία και για την ρήτρα της γεφύρωσης που συνδέει δηλαδή το κώδικα συνόρων Σέγγερ με το μηχανισμό της αξιολόγησης. Αυτές είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις κατά τη γνώμη μου. Και οι κόκκινε γραμμέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πέραν τούτου δεν μπορεί να ενδώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ελπίζω να δεχτεί το Συμβούλιο του όρου αυτού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συζητητές μας, τον κύριο Κοέλιο και την κυρία Βέμπερ, για την επιμονή τους και την αξιόλογη προσπάθειά τους στα δύο αυτά θέματα. Και όπως είπε ο κύριος Σεντσίου, θα ήθελα να υπενθυμίσω τις κόκκινες γραμμές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Μανσερβίση, εγώ δεν συμφωνώ με τη δική σας εκτίμηση ότι έχει σημειωθεί ένα μεγάλο βήμα πρόοδο. Είχαμε ε, αρκετές επαφές και διαπίστωσα το τελευταίο τριμερή διάλογο ήταν ελάχιστη η πρόοδος. Εμείς ε, οι πράσινοι επιμένουμε και στηρίζουμε περισσότερο την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επαναφορά του ελέγχου στα σύνορα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση όμως ε, του Συμβουλίου στο τελευταίο τριμερή διάλογο δείχνει ελάχιστη επιθυμία πρόοδου. Και εύλογα θέτει η κυρία Βέμπερ το ερώτημα. Μήπως ε, τελικά αντί να βελτιώσουμε τα πράγματα και να ενισχύσουμε ε, το Σέγγεν, θα επιδεινώσουμε τελικά την κατάσταση. Και όντως υπάρχει επιθυμία βελτίωσης. Ευχόμαστε ε, ολόθερμα καλή επιτυχία στην Κυπριακή Προεδρία αλλά με την παρούσα θέση του Συμβουλίου πολύ αφιβάλλουμε για την περαιτέρω πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Έρνστ. Εν τω μεταξύ, οι δύο εκθέσεις ε, ε, ε, κινούνται σε ονειρικό πεδίο. Στην αρχή είχαμε πει ότι δεν έχει νόημα σε όλη αυτή την υπόθεση και πιστεύουμε ότι οι ρυθμίσεις ουσιαστικά είναι καλές. Τώρα υπάρχει πόλεμος μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και κάπου ανάμεσα ενίκη Κομισιόν και αυτά που κρίνουμε θα πρέπει να τα αναγάγουμε στο ένα και μοναδικό ερώτημα. Πού το πάμε, τι επιδιώκουμε. Συμφωνήσαμε ότι όλα αυτά πρέπει να είναι κοινοτικές αποφάσεις όταν πρόκειται για επαναφορά ελέγχων συνόρων. Δεν γίνεται αυθαίρετα, για να αναφέρω το παράδειγμα της Δανίας εδώ. Όταν ακολουθήσουμε αυτό το στόχο λοιπόν, και αυτό ήταν ομόφωνη θέση στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν, τότε με το άρθρο 70 δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Όπως και να τα στρέψουμε και να τα γυρίσουμε τα πράγματα και όπως και να τα νοματίσουμε, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό το άρθρο δεν θα μας βοηθήσει και καμία κριτική δεν το στηρίζει. Μέχρι τώρα δεν προέκυψε τίποτε το ε, αξιόλογο και το χρήσιμο. Εμείς θέλουμε να πούμε το εξής. Εγώ είμαι κατοικός στα γερμανοτσεχικά σύνορα και τα λεωφορεία από την Τσεχία ελέγχονται και από την Πολωνία επίσης. κανένας στη χώρα αυτή δεν ε, πιστεύει ότι θα λειτουργήσει το άρθρο 70. Χρειάζονται αυστηρές ρυθμίσεις και υπ' αυτή την έννοια εμείς ό,τι υποβληθείτε είναι προτάσεις από το Συμβούλιο που θα τις πούμε συμβιβαστικές είτε οτιδήποτε άλλο θα τις κρίνουμε με αυστηρά κριτήρια γιατί γιατί όπως σας είπαμε πιστεύουμε ότι η, η, η σύσταση σίγουρα δεν εξυπηρετεί ούτε αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Έχουμε καθυστέρηση μεγάλη. Στις 5 θα έπρεπε να περάσουμε στο επόμενο θέμα ενώ είναι 5 και 4 οπότε το λογικό είναι να δώσουμε το λόγο στους εισηγητές να κλείσουν προσθέτοντας κάτι ακόμα, δεν χρειάζεται να μακρηγορήσουν, αλλά έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν ο καθένας τους δύο λόγια αν θέλουν. Ο κύριος Κοέλιο. Πρόεδρε, τα είπα όλα στην πρώτη μου παρέμβαση. Να προσθέσω κάποιο σχόλιο όμως θα ήθελα. Μία από τις διατάξεις που έχουμε στα νέα μέσα είναι η δυνατότητα οι ομάδες να πάνε σε εσωτερικά σύνορα και να διαπιστώσουν κατά πόσο υπάρχει έλεγχος παράνομος στα σύνορα ή ότι δεν υπάρχει. Σε αυτά τα σημεία του κειμένου, κατά την άποψή μου, προχωρούμε πιο πέρα από την τωρινή κατάσταση. Αν θέλουμε να δούμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία των νέων διατάξεων, με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ηγείται των ομάδων, με την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Υπάρχει δυνατότητα διαπίστωσης κατά πόσο γίνονται παράνομα. Με όλα αυτά μιλάμε ξεκάθαρα για καλές βελτιώσεις, για βελτιώσεις. Δεν κρύβω ότι υπάρχουν τα διαπιστωθέντα προβλήματα, αλλά αν μιλάμε για πρόοδο, έχουν επιτευχθεί αρκετές. Είναι μια καλή δυνατότητα Εάν μας δίνετε μια καλή δυνατότητα να καταφέρουμε να πετύχουμε συμβιβασμό, πρόεδρε να πω ότι μετά από συζήτηση με την Κυπριακή Προεδρία σήμερα συμφωνήσαμε ότι καταρχήν την Τρίτη θα γίνει και άλλος τριμερής διάλογος επικειμένου που θα μας υποβληθεί. Κάθε αξιολόγηση θα πρέπει να εδράζεται επικειμένων και θα δούμε τι θα γίνει από την Τρίτη και μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές που υπήρξαν συντομότατοι. Ευχαριστώ τον κύριο Ρασεβίση. δεν ξέρω αν θέλετε εν συντομία να προσθέσετε κάτι γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω. Αν επιτρέπετε να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Κοέλιο. Όχι μόνο αυτά που είπατε γίνατε. Κάποιος θα κάνει συγκεκριμένη πρόταση να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. και αυτό ακολουθεί την συνηθισμένη διαδικασία λήψης απόφασης. Άρα προσθέτουμε και κάτι πιο συγκεκριμένο, να γίνονται πράγματα, όχι απλώ να διαπιστώνται προβλήματα. Είναι ευαίσθητο το πλαίσιο βέβαια, αλλά απλώ ήθελα να ολοκληρώσω τα υποθέντα. Ευχαριστώ κύριε Μασαβίση. Θα τα ξαναπούμε σε επόμενη συνεδρίασή μα με το πακέτο για το άσυλο. Α προχωρήσουμε και α πάμε στο επόμενο σημείο της διάταξη. Προσοχή παρακαλώ περνάμε χωρίς άλλη καθυστέρηση στην κοινή συζήτηση των σημείων 6 και 7. Παρακαλώ. Επαναλαμβάνω. Θα έχουμε κοινή συζήτηση τώρα των σημείων 6 και 7. Αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξη Υπηκών Τρίτων Χωρών. Παρακαλώ ησυχία όσοι παραμείνετε στην αίθουσα και όσοι ε, φύγετε παρακαλώ επίσης ήσυχα. Και συζήτηση του σημείου 7 με θέμα την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για ορισμένα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες σε σχέση με την χρηματοοικονομική του σταθερότητα. Εισηγητής και για τα δύο θέματα είναι ο κύριος Νίλ Τόρβαλτς των Φιλελευθέρων. Θα ακούσουμε λοιπόν την παρουσίαση από τον εισηγητή μας, τον κύριο Τόρβαλτς και μετά θα δώσουμε το λόγο για σύντομο σχολιασμό στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Παρακαλώ χρόνου φίδου, γιατί έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να καλύψουμε το χρόνο που έχουμε χάσει. Ο κύριος Τόρβαλτς, ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω οι συνάδελφοι να έριξαν μια ματιά στα σχέδια εκθεσή μου, τουλάχιστον οι παρόντες. Εγώ συμφωνώ με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχήν γνωρίζουμε ότι ε, η οικονομική και η δημοσιονομική κρίση είχε σοβαρές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά των πολλών χωρομελών και επίσης ε, πηρέσει την ικανότητά τους ε, να τηρήσουν τις υποχρέωσεις χρηματοδότησης αυτών των τεσσάρων ταμείων στα πλαίσια του Γενικού Προγράμματος για την Αλληλεγγύη και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ωρών. Η διαχείριση το μεταναστευτικό ροών είναι σημαντικό θέμα για το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η ε, αδυναμία ενό κράτου μέλου να εξασφαλίσει σωστή διαχείριση και αποτελεσματική των μεταναστευτικών ροών επηρεάζει όχι μόνο την συγκεκριμένη χώρα, αλλά έχει επιπτώσει και σε όλε τις υπόλοιπε χώρε μέλη. Γι' αυτό είναι και προ όφελο όλων των χωρών μελών οι δεσμεύσει που έχουν αναλυθεί για την μετανάστευση να μην πληγούν από τι οικονομικέ δυσκολίε που αντιμετωπίζουν κάποιε χώρε μέλη. Και μάλιστα όσοι συμμετείχαν στην πρόσφατη αποστολή της Επιτροπής μας στην Ελλάδα διαπίστωσαν οι δύο ότι πολλά προγράμματα είναι αδύνατο να εφαρμοστούν χωρίς αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης. Για παράδειγμα, ανακαινήσεις των κέντρων κράτησης ή βελτίωση του τεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη διαχείριση των συνόρων οι χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ε, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο, στη χρηματοδότηση για τη σωστή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και εξαιτίας των σημαντικών αυτών οικονομικών δυσκολιών οι χώρες αυτές ε, αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ε, της συγχρηματοδότησης και τα προγράμματα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Δικαιολογείται λοιπόν αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης, γι' αυτό και συμφωνώ με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιτρέπει στα κράτη-μέλη που ζήτησαν ε, οικονομική αρρωγή να υποφεληθούν από αυτό το, την αύξηση. Ε, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Λετωνία και η Πορτογαλία είναι αυτές ε, οι έξι από τις 27 χώρες που υποφελούνται από, το, από την πρόταση αυτή που έχει στόχο να αυξήσει το ποσοστό στη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, μειώνοντας αντίστοιχα τις ανάγκες στη χρηματοδότησης ε, της ενδιαφερόμενης χώρας. Έτσι, το ποσοστό στη χρηματοδότηση θα ανέφθει στο 70% για σχέδια που αφορούν ειδικέ προτεραιότητε για όλα τα κράτη-μέρη που καλύπτονται από το Ταμείο Συνοχή ε, και αυξημένο δείκτη είναι το 95% κατά ανώτατο όριο. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο λόγο της ε, έκθεσή μου. Η μεταβολέ του δείκτη χρηματοδότηση των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν σοβαρέ δυσκολίε όσον αφορά τη δημοσιονομική του σταθερότητα δεν συνεπάγονται αύξηση των συνολικών ποσών για τα ελόγω ταμεία. Το συνολικό ετήσιο εθνικό κονδύλι που αφορά τι βασικέ πράξει θα παραμείνει αμετάβλητο, ενώ θα μειωθεί αντίστοιχα η εθνική συγχρηματοδότηση. Οπότε δεν θα υπάρξει καμία ε, οικονομική επίπτωση στη υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ε, ας μην ξεχνάμε και το θέμα τη συνοχή με τα άλλα κοινοτικά ταμεία. Αντίστοιχε αλλαγέ ε, στι απαιτήσει χρηματοδότηση έχουν ήδη εγκριθεί για τα, για τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχή, ε, το Ταμείο Γεωργική Ανάπτυξη και το Αλληλευτικό Ταμείο. Οπότε ε, μπορούμε να εφαρμόσουμε αντίστοιχε αυξήσει και στα ταμεία που διέπουν τις μεταναστευτικές ροές. Άλλωστε το μέτρο αυτό της αύξησης χρηματοδότησης είναι μόνο προσωρινό και δεν θα επηρεάσει την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Είναι σημαντική είναι σημασία ο αποτελεσματικό έλεγχο τη χρήση των πόρων και είναι κρίμα που η κατάχρηση, η κακή ε, απορρόφηση σε ορισμένα κράτη-μέλη επιδεινώνει την κατάσταση. Γι' αυτό και θα πρέπει να βελτιώσουμε τον έλεγχο και τις εξακριβώσεις ε, της διαχείρισης του συστήματος. Ε, και μάλιστα ο έλεγχος της διάμεσης αναθεώρησης είναι εξίσου απαραίτητος όσο και η συνεχής αποτελεσματική παρακολούθηση. Οπότε συνιστώ την έγκριση των δύο προτάσεων χωρίς τροπολογίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εγκρίνει τις προτάσεις χωρίς το δεοδο έλεγχο, αλλά υπό τις συνθήκες αυτές οι προτινόμενες αλλαγές είναι δικαιολογημένες και έχει ζωτική σημασία να εγκριθούν εντός του προτινόμενου χρονοδιαγράμματος, ώστε να έχουν πραγματικά τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε προγράμματα που χρήζουν χρηματοδότηση σε κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. Έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε ε, ομαλά αποφάσει για τα θέματα αυτά και ελπίζω να συμφωνήσουν και όλες οι πολιτικές ομάδες. Είμαι στη διάθεση των συναδέλφων για να απαντήσω σε απορίες τους ή να ακούσω τα σχόλιά τους. Πρώτα στον κύριο Αντουάν Σαββάρη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον εισηγητή για την έκθεσή του που υποστηρίζει πλήρω την πρόταση ευρωπαϊκή επιτροπή άνευ τροπολογιών. Δεν μπορούμε παρά να ε, εκφράσουμε την ευχαριστή μας για αυτή την ε, έκθεση και δεν έχουμε συμπληρωματικά σχόλια. Σα ευχαριστώ. Η Κυπριακή Προεδρία. Αργυρόπουλου. Κύριε Αργυρόπουλου. Exactly. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι συντομότατη κι εγώ. Θα βασίσω την παρέμβασή μου στην πρώτερη που έγινε στις 5 Νοεμβρίου. Ε, με τα χαρά σας ενημερώνουμε λέγοντας ότι περιμένουμε εντολή για να ξεκινήσει ο επίσημος τριμερής διάλογος με το Κοινοβούλιο περίπου μέσα Δεκεμβρίου θα λάβει χώρα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ξανά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για τη συνεργασία του και την καρποφόρα συνεργασία μέχρι τώρα, κυρίως από αυτού του χαρτοφυλακίου και προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία μαζί σας για την επίτευξη ταχεία συμφωνίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ας δούμε αν κάποια μέλη θέλουν το λόγο. Κύριε Πανικολάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για την εισαγωγή που μας έκανε και για την προσέγγιση που ακολούθησε αυτή η αλλαγή για τα Ταμείο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο ε, είναι μια προσαρμογή στην κρίση στην πραγματικότητα, αυτή η τροποποίηση και είναι μια ευρωπαϊκή αντίδραση ε, προς ε, βοήθεια των χωρών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ώστε να διατεθούν τα αναγκαία εργαλεία για την καταπολέμηση των κοινών ευρωπαϊκών προβλημάτων σε ένα περιβάλλον ε, πολύ μεγάλης κρίσης που πλήττει όλους αλλά κάποιες χώρες περισσότερο από άλλες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρξει συνοχή με, άλλες, ε, με άλλα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτές οι τροποποίησεις ήδη είχαν εφαρμοστεί στα διεθντικά ταμεία, ταμεία συνοχής. Ε, τα ανέφερε όλα ο εισηγητής. Όσον αφορά αυτά τα ζητήματα λοιπόν, όταν τα συζητάμε είναι πολύ σημαντικό να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη να κάνουν καλή χρήση της χρηματοδοτήσεως και βέβαια να χρησιμοποιηθούν καταρχήν αυτοί οι πόροι. Ακούσαμε την Επίτροπο την κυρία Μάστρομ η οποία μας είπε προηγουμένως ότι υπάρχουν χρήματα για τον τομέα αυτό, αλλά δυστυχώς ε, δεν υπάρχει επαρκές δυναμικό από πλευράς κρατών μελών για την χρήση τους. Καλωσορίζω λοιπόν την παρουσίαση που μας έκανε ο εισηγητής Ασκιώδης από το ΕΛΚ. Θα ακολουθήσω την προσέγγιση του. Δεν θα υποβάλω τροπολογίες ο ίδιος. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε και άλλες τροπολογίες από άλλους συναδέλφους της ομάδας μου. Θα διαβιβάσω αυτό το μήνυμα. Ήδη έχω κάνει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικό να μην χρονοτριβούμε διαπραγματευόμενοι σε συναντήσεις και τριμερείς διαλόγους αν μπορούμε να πετύχουμε τάχιστα αποτέλεσμα. Να ευχαριστήσω επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για τις θέσεις τους και βεβαίως για εκείνους που έχουν αμφιβολίες όσον αφορά αυτού του είδους τις ρυθμίσεις σε τέτοιες εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει να επενθυμίζουμε στον εαυτό μας κάθε φορά ότι παρόλο που αυξάνουμε τη συνεισφορά της Ευρώπης, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διεξάγεται ο πραγματικός έλεγχος και αξιολόγηση για τη χρήση των πόρων. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, πολλές ανάγκες, κυρίως για την Ελλάδα, τη χώρα μου. Υπενθυμίζω και την πρόσφατη αποστολή που πήγε στην Ελλάδα και όλοι οι συνάδελφοι είδαν τις ανάγκες που υπάρχουν ότι χρειάζεται στο μέτρο του δυνατού να Φόνται οι πόροι, οι ευρωπαϊκοί. Με αυτή την τροποποίηση δίνουμε ένα αποτελεσματικό εργαλείο και στις έξι χώρες, τις οποίες ανέφερε ο εισηγητής, και πιστεύω ότι αυτό θα μας δώσει καλά αποτελέσματα τον επόμενο χρόνο, όχι μόνο όσον αφορά την απορρόφηση της χρηματοδοτήσεως, αλλά και όσον αφορά θετικές πραγματικές εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου στις χώρες εκείνες που είναι στο επίκεντρο της οικονομικής αυτής κρίσης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Εν γέννη δεν βλέπουμε να υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε δεν θα έχουμε να υποβάλουμε και τροπολογίες για την ώρα. Έχω κάποιες ερωτήσει που απευθύνω προ εσά ή ίσως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ίσως αυτό με διαφωτίσει. Θα ήθελα να ξέρω ποια κράτη-μέλη θα ωφεληθούν πραγματικά από τα υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης, ακριβώς ποιε χώρες. Και πόσα χρήματα ε, δέχονται μέχρι τώρα πόσοι πόροι τους διατίθενται και πόσα χρήματα έχουν απορροφήσει μέχρι τώρα και πόσα έχουν ζητήσει. Ένα πρόβλημα με τα ταμεία αυτά δεν είναι μόνο τα ποσά που εμπεριέχουν. Η γραφειοκρατία όμως, ο ρυθμός απορρόφησης σε κάποιες χώρες είναι πρόβλημα όπως στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα εξασφαλίσει ότι η δυνατότητα απορρόφησης δεν αποτελεί πρόβλημα και ότι δεν υπάρχουν άλλα ε, ε, γραφειοκρατικά προβλήματα. οι γραφειοκρατικά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι χώρες που ζητούν αυτή την ενίσχυση. Όταν υπάρχει ποσοστό χρηματοδότησης 95% ή 100% τότε αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη ευθύνη ελέγχου πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σωστή χρήση των χρημάτων. Άρα και η ερώτηση. Εσείς πώς μπορείτε να είσαστε σίγουροι ότι μπορείτε να παίξετε σωστά τον ελεγκτικό σας ρόλο και ότι τα χρήματα θα δώσουν προς τη θέμενη αξία μέσω αποτελεσματικής χρήσεως. Το Ταμείο της Πρόσφυγες θα απορροφήσει πράγματι τα χρήματα που θα διτίθεται. Μια, ένας φορέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων έθεσε ερωτηματικά για πρώτερες δαπάνες στην Ελλάδα για το Ταμείο των Προσφύγων. Πώς είμαστε σίγουροι ότι τα χρήματα που διατίθεται φτάνουν πραγματικά στα χέρια των προσφύγων. η Κομισιόν. Γιατί έγιναν κάποιες παρατηρήσεις πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Τόρβα, τον εισηγητή μας. Ε, η κυρία Κέλλερ έκανε κάποια ε, θέματα, η Κομισιόν. Καλώς να απαντήσω σε ορισμένα θέματα, γιατί για τα άλλα θέλουμε πιο, πολλές, πιο πολλή ώρα για τις απαντήσεις. Ποιες είναι οι χώρες δικαιούχοι. Οι χώρες που θα υποφεληθούν από την αύξηση του ποστό χρηματοδότηση είναι η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η, η Ρουμανία, συγγνώμη, η Ισπανία μέσω του μηχανισμού ε, βοήθειας στο τραπεζικό σύστημα θα συμπεριληφθεί και στις επόμενες εβδομάδες και η Κύπρος. Αυτές είναι οι χώρες που θα υποφεληθούν από την αύξηση του ποστού χρηματοδότησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης. Η απόφαση αυτή ελήφθη κυρίως γιατί οι χώρες ε, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την κρατική χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν τα προγράμματα και τις δράσεις το θέμα της ε, απορρόφησης είναι δευτερεύον σε σχέση με τις ανησυχίες που αποτέλεσαν το γενεσιουργό λόγο της απόφασης. Η απόφαση αυτή θα επηρεάσει τα προγράμματα 2011, 2012 και 2013. Δεν έχουμε καμία ιδέα ήδη για το ποιο θα είναι το ποστό απορρόφησης. Υπάρχουν χώρες που έχουν πολλά, πολύ καλά ποστά απορρόφηση όπως η Ισπανία και... Από τις έξι αυτές χώρες δεν βλέπω χώρες που να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα απορρόφησης, με εξαίρεση την Ελλάδα ίσω. Το πρόβλημα όμως ε, της Ελλάδας ε, δεν έχει σχέση τόσο με αυτό το θέμα. Πάντως ε, η βάση της απόφασης είναι η ανάγκη αρρωγής προς τις χώρες αυτές για να συμπληρώσουν το ελληπές τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης και να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τα προγράμματα. Για το ιδιαίτερο ζήτημα του Ταμείου Προσφύγων δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν είμαι αρμόδιος για το θέμα αυτό θα διαβιβάσω στον αρμόδιο τον προβληματισμό σας και θα σας ε, στείλουμε γραπτός απάντηση. Επίσης, ε, αναφερθήκατε στην Ελλάδα. Έχει, έχουν θεσπιστεί πολλά μέτρα για να βοηθήσουμε την Ελλάδα προκειμένου να ενισχυθούν οι διοικητικές της ικανότητες. Μάλιστα ε, έχουμε θεσπίσει και μια task force σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικουρεί την Ελλάδα προκειμένου να πλουστευτούν οι διοικητικέ διαδικασίε και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα κονδύλια και τα ταμεία, να βελτιωθεί η ικανότητα των αρμοδίων αρχών να ε, υποβάλουν διαδικασίες ε, και διαγωνισμούς σε πιο σύντομες προθεσμίες γιατί ιδιαίτερα στο Ταμείο για τα Εξωτερικά Σύνορα αυτό είναι το πρόβλημα. Διαδικασίες ε, ε, διαγωνισμών και υποβολής προσφορών ε, με πιο μικρές προθεσμίες ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπει το Ταμείο. Και μια διευκρίνηση. Δεν θα αυξηθεί το συνολικό κονδύλιο της κάθε χώρας. Απλώς θα μειωθεί το ποσοστό χρηματοδότησης, αλλά δεν τροποποιείται ο προϋπολογισμός ε, ή το, ο προϋπολογισμός των ταμείων ε, ή το ετήσιο ποσοστό της κάθε χώρας, το ετήσιο κονδύλιο, συγγνώμη, της κάθε χώρας. Δεν ξέρω αν θέλετε να υποβάλλετε κάποιο σύντομο σχόλιο, αλλά μην επανέλθουμε στη συζήτηση, γιατί θα πρέπει να δευτερολογήσουν, να ο εισηγητής. Μα μιλούμε για το Ταμείο Προσφύγων. Έτσι δεν είναι. Α, για όλα τα ταμεία. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλούμε μόνο για το Ταμείο Προσφύγων και το Ταμείο ε, Εξωτερικών Συνόρων. Στην ε, αιτιολογική έκθεση αναφέρονται ρητά η Ουγγαρία και η Λετωνία. Αυτές οι χώρες δεν θα υποφεληθούν από την αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης, δεν θα λάβουν κονδύλια. δώστε απάντηση αν θέλετε, αλλά παρακαλώ επιγραμματικά γιατί έχουμε μείνει πίσω στο χρόνο. Όντως, το 2012 η Λετωνία δεν επωφελείται από το μηχανισμό αρρωγής, δεν θα ενταχθεί στο πρόγραμμα. Δεν θα υποβληθούν, δεν θα ληφθούν νέα κονδύλια. Δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται αύξηση του προϋπολογισμού του εθνικού ποσού για την κάθε χώρα, επαναλαμβάνω. Μόνο το ποσοστό χρηματοδότηση αυξάνεται. Yes, uh, just to... Ο εισηγητής. Ε, την πρώτη σας ερώτηση τη σκέφτηκα και εγώ και αυτό με προβλημάτισε όταν ε, πρωτοσχολήθηκα με το θέμα αυτό. Και δεν έχω τις απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα. Και τα κονδύλια για την εφαρμογή των προγραμμάτων μπορούμε να τα, μπορώ να σας τα δώσω πριν ψηφίσουμε, ώστε να έχουμε γνώση της κατάστασης. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο κέριο ερώτημα. Ευχαριστώ πάντως για τα σχόλιά σας και θα έχω επαφές με τους και Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε αυτό το ζήτημα σε χρόνο ρεκόρ τελικά. Ευχαριστώ τον εισηγητή και για τα σχολιά του, αλλά και για τις προσπάθειες ε, που κάνει. Ώστε να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα γρήγορα και να κερδίσουμε το χαμένο μας χρόνο. Μην ξεχνάτε και την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Λίγη στις 29 Νοεμβρίου. 29 Νοεμβρίου 2012 φυσικά, στις 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 17 ή 18 Δεκεμβρίου και στην Ολομέλεια προβλέπεται η ψηφοφορία τον επόμε... το Φεβρουάριο του επόμενου έτους, το Φεβρουάριο του 2013. Σας ευχαριστώ και περνάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης είναι έκθεση κυρίας Μακοβέη για τη δημιουργία του συστήματος Eurodac για τη σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Αναδιατύπωση. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε σήμερα τις τροπολογίες ε, για τον κανονισμό που προβλέπει σύσταση του συστήματος Eurodac. Στις 11 Οκτωβρίου είχαμε την πρώτη υποβολή της, του σχέδιου έκθεσης. Υποβλήθηκαν 162 τροπολογίες και στο μεταξύ προσθέθηκαν και άλλες 20, ε, 182 τελικά λοιπόν τροπολογίες έχουμε για την έκθεση αυτή. Θα ψηφίσουμε στις 17 ή 18 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή μας. Γι' αυτό και θα ακούσουμε τώρα το σχολιασμό των τροπολογιών από την εισηγητριά μας, την κυρία Μακοβέη και μιας θα ακολουθεί συζήτηση. Παρακαλώ κυρία Μακοβέη, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ. Η Eurodac ε, με βάση αρνητικές ή θετικές απαντήσεις ε, είναι μέρος του πακέτου, πακέτου που θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012. Η θέση του ΕΛΚ είναι να διατηρηθεί το πακέτο και ταυτόχρονα να ψηφιστεί στην Ολομέλεια ε, μαζί με την οδηγία για τις διαδικασίες και το Eurodac. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για το ενδιαφέρον που έδειξαν και για τις πολυάριθμες τροπολογίες. Τώρα, για τις τροπολογίες. Κάποιες από αυτές δίνουν περισσότερες διασφαλίσεις ε, για την άσκηση της επιβολής του νόμου και την πρόσβαση ε, και, τη, αυτών, και της ε, Europol στη βάση δεδομένων. θα τις δεχτώ αν δεν αποκλείουν τη διαδικασία, δεν την καθιστούν αδύνατη. Θα σας δείξω κάποιες, κάποια παραδείγματα τροπολογιών που μπορώ να υποστηρίξω για την ανεξαρτησία της αρχής επαλήθευσης της, ε, των ε, αρχών που, ε, στους οποίους έχει γίνει η ανάθεση το σύστημα πριν ζητηθούν για αντιπαραβολή στο Eurodac ή όταν υπάρχουν έγκυρες υποψίες ότι ποιος έχει διαπράξει ε, μια αξιόπινη πράξη, έχει ζητήσει διεθνή προστασία και ε, εδώ πρέπει να υπάρχει πρόσβαση της ε, Europol στη βάση δεδομένων. Τώρα, ε, ό,τι αφορά το, την, κατάργηση του συστήματος πάνω στη βάση hit-no-hit, no hit, θετική ή αρνητική απάντηση ή καμία απάντηση, ε, αυτά είπα να τα διαγράψουμε. Ε, επίσης είμαι διατεθειμένη να συζητήσω συμβιβαστικέ τροπολογίες. Ε, ενημέρωσα τη γραμματεία και νομίζω, ελπίζω να συνταχθούν πριν από τη συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές την ερχόμενη Πέμπτη. Θα έλεγα τέλος ότι ελπίζω ότι θα έχουμε γόνιμη συζήτηση ε, όταν μιλήσουμε για τους φακέλους αυτούς και θα τηρηθούν οι δεσμεύσει σε σχέση με το πακέτο άσυλο και θα επιδειχθεί η αλληλεγγύη με βάση ενιαίο καθεστώς ε, ανθρώπων που ζήτησαν διεθνή προστασία. Που, που τους δόθηκε ε, διεθνής προστα... προστασίας. Λοιπόν, θέλω να ξαναπώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο αν θέλω να πάρω το λόγο σε αυτό το στάδιο των συζητήσεων. Έχετε το λόγο, κυρία μου. Η Κομισιόν ε, υπέβαλε την πρόταση για να υπάρχει πρόσβαση ε, από τις διοικητικές αρχές ε, για να διασφαλιστεί ότι η ακαιρεότητα του συστήματος ασύλου θα διατηρηθεί. Ε, κατά συνέπεια ε, ε, είδαμε πολλές τροπολογίες για πρακτικές διασφαλίσεις που προστατεύουν τους ετούντες άσυλο και η Κομισιόν είναι ανοιχτή σε πολλές προτάσεις που έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζουμε ότι το συμβιβαστικό κείμενο δεν θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί ενσωματώνοντας κάποιες τροπολογίες των βουλευτών και μαζί με κάποιες τροπολογίες που έχουν συμφωνηθεί από το Συμβούλιο ε, με βάση την εντολή της Κορεπέρ στις 10 ε, Οκτωβρίου. Κάποια παραδείγματα. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για τον κανονισμό Eurodac κάθε φορά που λαμβάνουν τα αποτυπώματα. Δεν θα τους λέμε μόνο για το κανονισμό Δουβλίνου, αλλά και τη δυνατότητα ιδιοκτικές αρχές ε, να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους αυτά. Για παράδειγμα, η 139 τροπολογία είναι αποδεκτή από εμάς. Παράλληλα, ε, βεβαίως θέλουμε πάρα πολύ να διασφαλιστεί ότι το κείμενο θα ε, μας αφήσει με ένα λειτουργικό σύστημα Eurodac και σε σχέση με τις ε, τακτικές ε, επιχειρήσεις που στηρίζουν τον κανονισμό του Δουβλίνου και την πρόσβαση από τις διοκτικές αρχές. Έτσι υπάρχουν προτινόμενες τροπολογίες όπου δείχνουμε κατανόηση το πνεύμα που διέπει τη διατύπωση, αλλά θέλουμε να δουλέψουμε περισσότερο με τους βουλευτές για να ε, δούμε μήπως μπορούν να τροποποιηθούν λίγο οι τροπολογίες ούτως ώστε να συνάδουν με το συνολικό στόχο που είναι να έχουμε στο τέλος λειτουργικό σύστημα Eurodac. Μια τρίτη κατηγορία τροπολογιών μας φαίνεται ότι βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού, για παράδειγμα η 93 και 94 για το αποτέλεσμα ε, για μια αίτηση ασύλου στην περίπτωση που έχουν καταστραφεί τα δακτυλικά αποτυπώματα και δεν μπορούν έτσι τα δεδομένα να σταλούν στο Eurodac, δεν αντίκουν στον κανονισμό. Εκεί θα μιλήσουμε για την οδηγία για, ο, για τους ζητούντες άσυλο. Επίσης η 148 για την χρηματοδότηση και τη στελέχωση για την, ε, τις εποπτικές αρχές. Πιστεύουμε ότι και αυτή είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του κανονισμού Eurodac και δεν είναι παραδεκτή τροπολογία. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, να πω ότι βεβαίως ελπίζουμε ότι οι βουλευτές που ε, ζητούν ε, πρόσβαση από τις διεκτικές αρχές στο Eurodac ε, το θεωρούν σημαντικό, είναι σημαντική εξέλιξη. Ε, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τα αξιότιμα μέλη όμως να μην ακολουθήσουν ε, την οδό της ε, αποκλεισμού της πρόσβασης για να ολοκληρωθεί βραχυπρόθεσμα το σύστημα ασύλου και δεύτερον και πιο σημαντικά γιατί υπάρχει ανάγκη να κλείσει το κενό ενημέρωσης που αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών αυτή την κατηγορία για να ε, ε, εντοπιστούν πράξεις ε, τρομοκρατίας ή σοβαρού εγκλήματος. Ήδη σε προηγούμενες συνεδριάσεις θα έχουμε πει αυτά. Τέλος, να επαναλάβω ότι είμαστε ανοιχτοί σε μελλοντική στενή συνεργασία με τα αξιότιμα μέλη για να βρούμε έναν κατάλληλο συμβιβασμό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ωραία, τώρα να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Προεδρίας, τον κύριο Παπαγεωργίου. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για το λόγο και ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία που έχουμε στα πλαίσια του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Το Συμβούλιο εξέτασε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιστεύει ότι με σύντομες και γόνιμες διαπραγματεύσεις θα καταλήξουμε σε συμφωνία μεταξύ των δύο σχελών της νομοθετικής αρχής πιστεύω ότι μπορούμε να ομαδοποιήσουμε σε τρεις κατηγορίες τις τροπολογίες αυτές που θέλουν να ε, διαγράψουν την πρόσβαση των διοκτικών αρχών στις ε, πληροφορίες ή να την παρακολύσουν ε, καθιστώντας ανέφεκτη, κάτι που είναι ασύμβατο με τις θέσεις του Συμβουλίου και θα χαρούμε αν οι ευρωβουλευτές καταβάλουν μια προσπάθεια και καταψηφίσουν τελικά και την κατηγορία αυτών των τροπολογιών. Η δεύτερη κατηγορία τροπολογιών ε, ενισχύει τις εγγύησεις ε, πρόσβασης ε, των αρχών επιβολής του νόμου, των δεκτικών αρχών. Κατά τη γνώμη μου, τέτοιες τροπολογίες αποτελούν απαραίτητο στοιχείο του τριμερούς διαλόγου και θεωρούμε ότι θα είναι εύκολη η συμφωνία στους, των, στις τροπολογίες αυτές. Και η τρίτη κατηγορία τροπολογιών αφορά τις τεχνικές τροπολογίες. Σε πολλές περιπτώσεις ήδη καλύφθηκαν από το κείμενο του Συμβουλίου, που είναι μεταγενέστερο από το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο εσείς στηριχθήκατε. Θεωρούμε ότι εύκολα μπορούν να διαθετηθούν σε τεχνικό επίπεδο και να επισημάνω ότι η ημερομηνία για τον ε, διάλογο για τη συζήτηση ανατολισμού στη ΛΥΜΠΕ θα ακυρώσει τις προσπάθειες διεκπαιρέωσης ε, των ε, ε, διαπραγματεύσεων της αναδιατύπωσης μέχρι τα τέλη του έτους και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να καταβάλουμε προσπάθεια στα πλαίσια της εμβέσης εμπιστοσύνη να διεκπαιρεώσουμε το συντομότερο δυνατό τα θέματα αυτά. Φυσικά λαμβάνουμε υπόψη τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την σημαντική πρόοδο που σημειώσαμε στα άλλα ζητήματα. Οπότε εξηγήσαμε τις, σας εξηγήσαμε τις δυσκολίες μας, κύριε Πρόεδρε, και τις διαβιβάσαμε και στην εισηγήτρια. Το Συμβούλιο θα εκτιμήσει ιδιαίτερως ε, τις προσπάθειες ε, της ΛΥΜΠΕ και τη δυνατότητα ε, διοργάνωση έκτακτης συνεδρίασης ε, για την συζήτηση ανατολισμού, ίσως και στην Ολομέλεια, την επόμενη Ολομέλεια του Στρασβούργου, ώστε να ξεκινήσουν ε, πάρα αυτά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των συνομοθετών, προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία εντός των χρονικών ορίων. Γνωρίζουμε βέβαια ότι ίσως ανακύψουν κάποια πρακτικά ζητήματα ως προς την ε, ημερομηνία της συνεδρίας, αλλά πιστεύουμε ότι χρειάζεται καλή βούληση και από τα διαθεσμικά όργανα, προκειμένου να θεσπιστεί εντός των χρονικών ορίων το νομικό πλαίσιο που χρειαζόμαστε. Καλώς, έχω ένα κατάλογο των ομιλητών. Κυρία Ζίμπελ πρώτα. Thank you, Mr. President. Unfortunately, our... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς ε, ο συνάδελφος Κλοντ Μπεράς που είναι αρμόδιος για το θέμα αυτό δεν ε, ε, μπόρεσε να έρθει. Θα σας ενημερώσω εγώ για τη θέση των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Καταρχήν να ξεκινήσουμε τις διάφορες τροπολογίες. Φάνηκε με αυτέ ότι η επιμονή μας ε, για ένα πιο παρατεταμένο χρονοδιάγραμμα από το αρχικά προβλεπόμενο ήταν απαραίτητη. Δεν, θα, θέλουμε τεχνικώς να παρελκύσουμε, να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία, αλλά να ε, επιτρέψουμε στο Κοινοβούλιο τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθεί με το σημαντικό αυτό το θέμα. Θέλουμε τον απαραίτητο χρόνο για να εξετάσουμε ένα ζήτημα και μια έκθεση που θα έχει μεγάλες επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα. Από τις τροπολογίες είναι σαφές και εμφανές ότι έχουμε σοβαρές ανησυχίες τουλάχιστον για ένα θέμα που αφορά την πρόσβαση των διοκτικών αρχών στη Eurodac και των οργάνων επιβολής του νόμου. Βέβαια, αν η πρόσβαση των διεκτικών αρχών επιτραπεί στα στοιχεία της Eurodac, έχουμε και κάποιες ε, πλέον ανησυχίες. Μερικές ήδη αναφέρθηκαν, εγώ θα επικεντρωθώ ε, στο θέμα των ε, στην διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτες χώρες και των δακτυλικών αποτυπωμάτων και φυσικά στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων, γιατί τι θα γίνει με τα στοιχεία τους. Αυτά τα σημεία φυσικά είναι ενδεικτικά. Έχουμε και άλλες ανησυχίες. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες των άλλων ομάδων, είναι σαφές ότι υπάρχει δυνατότητα κατάληξη συμβαστικές τροπολογίες και ευελπιστώ ότι θα καταβάλει σχετικέ προσπάθειες η συγκεντρία. Τώρα επανέρχομαι στο πρώτο μου σχόλιο. Το χρονοδιάγραμμα. Οι συντονιστέ τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών συμφώνησαν στο χρονοδιάγραμμα που θα υποστηρίξει και η δική μα ομάδα μου όλη αυτή τη βδομάδα έχουμε τις συνεδρίες των σκιωδών εισηγητών. Μία συντμίση του χρονοδιαγράμματος δεν θα μας ε, επιτρέψει να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Κέλλερ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Yes. If I can have uh, kind attention. Um, so, we already expressed. Ήδη εκφράσαμε τις γενικά τις ανησυχίες μας επανειλημμένα. Δεν θα χάσω την ευκαιρία να πω ότι η αναλογικότητα και αναγκαιότητα αυτού του άξονα της επιβολής του νόμου δεν ε, δικαιολογούνται με κάποιο τρόπο. Δεν είναι δική μου άποψη. Ο Ευρωπαϊκός Ελεγκτής ε, Επόπτης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων το είπε και είπατε αρμοστία το για τους ε, πρόσφυγες. Τονίζει ότι η αναλογικότητα, η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα της προτάσεως για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκλημάτων πρέπει να εξεταστεί και να επιβεβαιωθεί πριν συμφωνηθεί ε, και συμφωνώ με αυτή τη δήλωση. Και είπατε αρμοστία επίσης αναφέρει και πολλές άλλες συστάσεις και αναφέρει και τη δυνατότητα να στιγματιστούν οι ετούντε άσυλο που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα και επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αμφιβολίες περί αυτού θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η αρμοστία έχει κάποια εμπειρία όσον αφορά την προστασία των προσφύγων και την προστασία των ετούντων άσυλο. Και ίσω έπρεπε να το λάβουν υπόψη. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι επιθυμεί να ενημερώνει τους ανθρώπους αυτούς των οποίων τα στοιχεία από το αντικείμενο επεξεργασία για το τι γίνεται. Τι γίνεται με αυτούς που είναι ήδη στη βάση δεδομένων. Δεν θα ενημερωθούν γι' αυτό ότι χρησιμοποιούν τα στοιχεία τους για εντελώς διαφορετικούς σκοπούς από ότι όταν δώσαν τα στοιχεία τους αρχικά. Και αυτό είναι σαφής παραβίαση κάθε αρχής προστασίας των δεδομένων. Η Αρμοστία αναφέρει επίσης ότι ότι μπορούν να δοθούν τα στοιχεία μετά από κάποιο πλήγμα σε τρίτη χώρα, μετά από ένα hit μάλλον, μπορούν να δοθούν σε τρίτη χώρα. Δεν υπάρχει συμφωνία με τις τρίτες χώρες όσον αφορά το τι γίνονται αυτά τα στοιχεία. Δεν καταλήξαμε σε κάποια λύση. Ασχολούμαστε με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αυτό το θέμα δεν το λύνει. Η Προεδρία είπε ότι θα είναι δύσκολο να τελειώσει το σύστημα ασύλου μέχρι το θέτους αν δεν βιαστούμε. Η Επίτροπο Μάλστρομ έκανε δηλώσει στι εφημερίδε και έλεγε ότι πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, νομίζω ότι αυτή το είπε, αν θυμάμαι σωστά, είμαι αρκετά σίγουρη ότι το είπε, ότι το σύστημα ασύλου θα είναι ε, έτοιμο το νωρίτερο τον Ιανουάριο. Από πού προέρχονται αυτέ οι δύο διαφορετικέ απόψει. Και τέλο, προ την κυρία Μακοβέ, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν Είναι ανοιχτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεγαλύτερες ρήτρες διαφύλαξης. Ίσως μπορούμε να συμβαστούμε εκεί. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Έχουμε συνάντηση σχεδόν την Πέμπτη. Δεν ξέρω πώ κινείστε εσεί. Εγώ πρέπει να είμαι στην εκλογική μου περιφέρεια την Πέμπτη. Και πιθανότατα οι περισσότεροι από εσά. Άρα δεν είναι δυνατόν να αλλάξω το πρόγραμμά μου και να απογοητεύσω του πολίτε ε, και να πάω από Δευτέρα στην Πέμπτη. Λοιπόν, Τετάρτη το απόγευμα θα έπραγουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Οι τροπολογίες μας επί μακρόν βρίσκονται εκεί. Και για να υπάρχουν σωστές συμβαστικές πρέπει να συζητηθούν και όχι την τελευταία στιγμή. Αυτά είχα να πω. Σας παρακαλώ εξετάστε κατά πόσο θέλετε να βελτιώσετε αυτό το κείμενο που θέτει ένα αμφιβόλο την πολιτική μας την προστασία των δεδομένων που αμφισβητεί και θέτει ένα αμφιβόλωτο το πώς αντιμετωπίζουμε τι ετούντες άσυλο, πώς αντιμετωπίζουμε τις άκρως ευάλωτες ομάδες και δεν δίνεται απάντηση στο ερώτημα πώς θα αποφύγουμε και άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις μέσω αυτής της πρόσβασης σε πάρα πολύ ευαίσθητε βάσει δεδομένων. Ευχαριστώ. Εκτό αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στάνεται την υποχρέωση. Ε, κύριε Τόρβαλτς, ναι. Το πρόβλημα είναι ότι η Σάρα Λάλτφορ δεν αισθάνεται πολύ καλά σήμερα. Οπότε, όπως βλέπετε, δεν ήρθε. Και πολλοί άλλοι φαίνεται ότι αισθάνονται ασχημούτσικα. Τέλο πάντων, δεν δίθεται αυτό το θέμα. Έχω κάποιε δικέ παρατηρήσει να σα διαβιβάσω. Δεν συμφωνώ με αυτά που διαβάσω. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για το έργο που κάνει για αυτό το θέμα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε τελικό αποτέλεσμα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ε, σε μερικέ εβδομάδε και γρήγορη έγκριση στην Ολομέλεια. Δεν έχω πρόβλημα όσον αφορά τι τροπολογίε, τη εισηγήτρια εκτό από την 11 και 14 που δεν βλέπω λόγο να αλλάξουμε τα στατιστικά στοιχεία κάθε μήνα και ούτε έχει αντίρρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Αλλά τροπολογίε που έχουν στόχο την ενίσχυση προστασία των ατόμων και την οδηγία και να υπάρχει συγκεκριμένο σκοπό των στοιχείων. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερα μέτρα προστασίας από ό,τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είναι αποδεκτό το μέτρο. Συμφωνώ με του συναδέλφους που ζητούν το Eurodac να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχουν ε, λογική, λογικά αίτια να θεωρούν ότι ο, κάποιος που έχει διαπράξει ένα έγκλημα ζητά διεθνή προστασία. Θα και αυτοί που συλλαμβάνονται στα σύνορα και αυτοί που βρίσκεται ότι ε, διαμένουν παράνομα εντός των κρατών μελών ε, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για αυτούς. Για να είναι ανάλογη η χρήση του Eurodac πρέπει να έχει λόγους να πιστεύει η αστυνομία ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία για συγκεκριμένη έρευνα και ότι η χρήση των στοιχείων συμβάλλει στην επιτυχή διελεύκανση της υποθέσεως. Ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια και όλες οι διαθέσιμες βάσεις ε, δεδομένων δεν αρκούν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ευάλωτοι και πολύ συχνά στιγματίζονται και είναι αντικείμενα διακριτική μεταχείριση σε κάποια κατημέλη. Αυτό που να το αποφύγουμε. Κάποιοι λένε ότι δεν θα κάνει διαφορά γιατί τα κράτη-μέλη του ή άλλω ε, εξετάζουν αυτέ τι βάσει δεδομένων του και συνεργάζονται με τα άλλα κράτη-μέλη όσον αφορά του ε, και χρησιμοποιούν τα στοιχεία για του ετούντε άσυλο Πρέπει όμως το Κοινοβούλιο να φροντίσει να θεσπίζεται νομοθεσία που συμφωνεί με τις αρχές μας. Το ότι υπάρχουν αυτέ οι πρακτικέ ήδη σε κάποια κράτη-μέλη που παραβιάζουν του κανόνε σημαίνει ότι πρέπει να θεσπίζουμε κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντιθέτω, μπορούμε να εμπνεύσουμε του νομοθέτε των κρατών μελών να θεσπίσουν σωστή νομοθεσία και ζητώ και συγγνώμη από του διερμηνεί που ήμουν πολύ γρήγορο. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο, κύριε Δεν ξέρω, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θέλει οπωσδήποτε να κάνει ένα σχόλιο πριν ξαναδώσουμε το λόγο στην εισηγήτριά μας την κυρία Μακοβέη. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Ναι, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλω κάποιο σχόλιο. Καταρχήν, η πρόσβαση των δικτικών αρχών είναι ο στόχο του προγράμματος. Δεν μπορούμε να δεχτούμε, είναι αδύνατο να δεχτούμε τροπολογίε που παρεμποδίζουν αυτή την πρόσβαση των διεκτικών αρχών στα στοιχεία της Eurodac. Τώρα, ε, είναι σημαντικό και το θέμα της χρήσης των δακτυλικών ε, αποτυπωμάτων στην, ε, στο χώρο του εγκλήματος και δεν μπορούμε να δεχτούμε τις ε, τροπολογίες που καθιστούν ανέφικτη μια τέτοια χρήση. Σε ό,τι αφορά την αναλογικότητα, το σχόλιο της κυρίας Κέλλερ. Μα περί αυτού πρόκειται κυρία Κέλλερ. Θέλουμε να δούμε τι είναι αναλογικό εδώ. Έχουμε αφενό ε, την ανάγκη καταπολέμησης ε, σοβαρών αξιόπινων πράξεων και τρομοκρατία, μόνο τέτοιων πράξεων και αφετέρου έχουμε πρόσβαση των διεκτικών αρχών. Εμεί ε, επανειλημμένω είπαμε ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλουμε αυτό το σύστημα να γίνει όσο πιο στεγανό γίνεται σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και επαναλαμβάνω το εχέγγυο ότι είναι έσχατη η λύση πρόσβαση των διεκτικών αρχών και δεν γίνονται αλληστηματικοί έλεγχοι ε, και απαγορεύεται η διαβίβαση τέτοιων δεδομένων σε τρίτες χώρες. Έχουμε αυτό το σύστημα hit or για να περιορίσουμε την ε, ανταλλαγή δεδομένων όσο γίνεται. Και μην ξεχνάτε ότι ήδη σήμερα είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των χωρών μελών. Αυτό που κάνουμε εδώ με τη συγκεκριμένη πρόταση είναι να θεσπίσουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, ενισχύοντας μάλιστα την προστασία των δεδομένων, προσθέτοντας και νέα εχέγγυα είναι πολύ καλύτερο από ότι να γίνεται διμερό μεταξύ των κρατών μελών αυτή η ανταλλαγή. Ελπίζουμε η πρόταση αυτή να ε, διεκπαιρεωθεί το συντομότερο δυνατό και μακάρι μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου όπως ε, εύχεται το Συμβούλιο, αλλά έστω και τον Ιανουάριο δεν, έχει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά το ότι στιγματίζονται οι αιτούντες στο άσυλο, θα το εξετάσουμε και αυτό στις ε, διάφορες συναντήσεις. Αλλά μην ξεχνάτε ότι η πρόταση για αξιολόγηση, για διάμεση αξιολόγηση μετά από κάποιο χρόνο εφαρμογής επίσης ε, προβλέπεται. Άλλωστε, άλλωστε ε, προσπαθούμε να αποφύγω αυτό το θέμα, να στιγματιστούν οι έτοντες άσυλο από τις διοκτικέ αρχές. Ευχαριστώ από αυτά προς το παρόν. Η συγκέντρια. εν συντομία, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο στη νέα πρόταση. Έχουμε δύο χρόνια που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και μάλιστα ήταν ε, και όμοιρος η πρόταση αυτή ε, για την συζήτηση άλλων παρεφερών θεμάτων. Πάντως, ε, εγώ ελπίζω ότι θα καταφέρουμε έστω και τον Ιανουάριο να προωθήσουμε και τις προτάσεις για το Δουβλίνο και την πρόταση για την Eurodac. Δύο φορέ συναντήθηκα με του κοιόδη εξετάσαμε το θέμα του χρονοδιαγράμματο, ακούσαμε τι παρουσιάσει του Συμβουλίου, τη Επιτροπή και η Επιτροπή έδωσε κάποιες απαντήσεις για το πώς θα εφαρμοστεί εμπράκτος αυτό το θέμα χρειαζόμαστε μια ισορροπία. Και εγώ είμαι υπέρ αυτής της ισορροπίας μεταξύ αφενός της ανάγκης να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και τα σοβαρά εγκλήματα και αφετέρου της ανάγκης να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων και ιδιαίτερα να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Θα πρέπει λοιπόν η ισορροπία να είναι το ζητούμενο και να μην κλείνουμε προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Υπάρχουν πολλέ δικλείδες προστασία και πολλά εχέγγυα στην πρόταση αυτή και από τις τροπολογίες θα δεχτώ όσες ε, δεν ε, ε, παρεμποδίζουν τη διαδικασία αυτή αλλά όσες την ευνοούν. Και χαίρομαι που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε την ίδια θέση. Υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βλέπω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ της πρότασης του Συμβουλίου να ψηφίσουμε λίγο νωρίτερα δεν είναι καινούριο το θέμα, μας απασχολεί εδώ και δύο χρόνια και όλα τα ζητήματα αναλύθηκαν διεξοδικά σε αυτή τη διετία. Και για τη συνεδρία των σχεδόν εισηγητών που προγραμματίστηκε για την Πέμπτη. Λυπάμαι δεν ευκαιρούν όλοι οι συνάδελφοι ε, και δεν θα έρθουν. Και εγώ αγκάστηκα να αναβάλω το ταξίδι μου σε εκλογική μου περιφέρεια για να είμαι παρούσα στη συνεδρίαση. Θα σας στείλω το συντομότερο δυνατό τις συμβαστικές τροπολογίες στα αγγλικά και ελπίζω να συμφωνείτε να τις εξετάσετε στα αγγλικά, τις συμβαστικές τουλάχιστον τροπολογίες. Καλώς. Ακούσαμε λοιπόν και πάλι την εισηγητριά μας την κυρία Μακοβέ και μην ξεχνάτε ότι η ψηφοφορία για το σημείο αυτό θα γίνει στη συνεδρίαση της 17ης ή 18ης Δεκεμβρίου. Οπότε, αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, μπορούμε να προχωρήσουμε στο τελευταίο σημείο της απογευματινής μας σημερινής διάταξης, το σημείο 9 δηλαδή, που αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαδικασία χορήγησης και ανκλήσης της διεθνούς προστασίας στα κράτη-μέλη. Αναδιατύπωση. Η συγγήτριά μας είναι η κυρία Σιλβίκη Γιώμ. Θα ακούσουμε πρώτα τα δικά τα σχόλια, δικά της σχόλια για την οδηγία που αφορά τις διαδικασίες ασύλου και θα μας παρουσιάσει την πρόοδο των τριμερών διαπραγματεύσεων που ήταν τρεις στον αριθμό μέχρι στιγμής. Κατόπιν θα ακούσουμε το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ολοκληρώσουμε την απογευματινή μα συνεδρίαση. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε αργότερα και μια άτυπη ομάδα εργασία ακριβώ για το πακέτο του ασύλου. Ευχαριστώ. Πάμε και πιο γρήγορα μάλιστα. Πρόκειται περί ενημέρωσης που δίνω στους συναδέλφους, αυτούς που είναι παρόντες τουλάχιστον. Αυτά που θα πω δεν θα εκπλήσουν το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάναμε κάποιες πρόοδους όσον αφορά την ε, οδηγία να πω κάτι που είναι σωστό. Αυτό το κείμενο είναι περιπλοκότατο, μακροσκελέστατο και πρέπει να χαρούμε διότι προχωρήσαν οι συζητήσεις. Είμαι σίγουρο ότι θα κατορθώσουμε να βρούμε ικανοποιητική λύση και τα τρία θεσμικά όργανα επί πολυαρίθμων σημείων, ακόμα και αν αναφέρω αυτά τα σημεία που είναι προβληματικά πρόγραμμα. Έχουν προγραμματιστεί δύο τριμερείς διάλογοι. Θα είμαστε στον πέμπτο και 4 Δεκεμβρίου θα γίνει και ο έκτος. Και αν εδώ και αρκετό καιρό έχω πάψει να πιστεύω στον Άγιο Βασίλη, ελπίζω ότι ο έκτος αυτός τριμερής διάλογος μπορεί να οδηγήσει αποτέλεσμα. Αλλά για να γίνει αυτό ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι μέσα στην τελική ευθεία το Συμβούλιο. Και ισχύει αυτό που είπα ο συναδέλφος ότι το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης πλήρης και ότι το Κοινοβούλιο έχει και αυτό τις ερυθρές γραμμές, τις κόκκινες γραμμές και τις φιλοδοξίες του. Γι' αυτό θέλω να επενθυμίσω εν συντομία την ακολουθησή σα προσέγγιση Πλευράς Κοινοβουλίου από όταν ξεκίνησε συζητήσεις. Τρία σημεία θέσαμε στοιχείο. Πρώτα απ' όλα θέλαμε γενική ισορροπία αυτή θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε εναρμονισμένες, δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες. Και για να στηρίξουμε αυτή την στρατηγική, ακολουθήσαμε τέσσερις άξονες. Το δίκαιο, αποτελεσματικότητα, ποιότητα και αξιολόγηση. Και για κάθε άξονα ε, θέλαμε σαν κοινοβούλιο να ξέρει ότι έχουμε γενική ισορροπία μετά τη συζήτηση στοιχεία που κερδίσαμε, αλλά και διατάξεις που χάσαμε, αλλά γενικά να επικρατεί μια ισορροπία. Δεν μπορούμε να εστιαζόμεθα επί μια συγκεκριμένη διατάξεω. Πρέπει να εξετάσουμε ολιστικά το κείμενο. και να βελτιώσουμε ε, κάποιες λεπτομέρειες της διατάξης. Αυτό δεν, αυτά δεν αποκλείουν σαφή δήλωση θέσεων του Κοινοβουλίου. Φτάσαμε στα όρια μας και στις απογοητεύσεις. Και όταν χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Όπως έλεγα θέλαμε γενική ισορροπία. Αυτό προσπαθούμε σταδιακά να πετύχουμε. Στον τελευταίο τριμερή διάλογο εκμεταλλεύτηκε πλήρως το Κοινοβούλιο τα περιθώρια λιγμών που είχε. Πρέπει να αναφέρω τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε. Πρώτο σημείο το θέμα της κατάρτισης του προσωπικού του αρμοδίου και το Κοινοβούλιο επέμενε επί της κατάρτισης του προσωπικού των άλλων αρμοδίων αρχών. Δεν θα επισέδω σε λεπτομέρειες του κειμένου, που είναι περιπλοκότατο όπως σας είπα. Το θέμα της εκπαίδευσης κατά της επαρκούς για μας είναι σημαντικότατο. Και ξέρω ότι δεν είναι σημαντικό μόνο για μας. Δεύτερο σημείο, καλύτερη πλαισίωση των διατάξεων Κάτι που επιτρέπει στα κράτη-μέλη την ολοκλήρωση της διαδικασίας να την αναβάλουν αν επικρατεί κάποια βεβαιότητα στη χώρα καταγωγής του ετούντος. Και αυτό το θέμα, η αβεβαιότητα και τι πλαισίωση απαιτεί είναι κάτι που είναι σημαντικό για μας. Τρίτο, η καταχώρηση, η καταγραφή της συνέντευξης. Λέγαμε ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό αυτό αν η αρχή που καθορίζει ε, αποφασίζει να υπάρξει αυτή η καταγραφή και ποιες οι σημαντικές εξαιρέσεις σε κάποιες διαδικασίες. Κυρίως τους μη συνοδευόμενους ανηλίκους και τα ευάλωτα άτομα και εκείνα τα άτομα που έχουν ιδιαίτερες διαδικαστικές ανάγκες. Είναι δύσκολα σημεία, δεν είναι καινοτομία αυτή για το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά τα σημεία επεξεργαζόμαστε Θέλουμε να ακολουθήσουμε, όπως σας είπα, ρεαλιστική, ε, λογική προσέγγιση. Θέλαμε γενική ισορροπία. Αυτή είναι η του Κοινοβουλίου και θα θέλαμε να ληφθεί υπόψη. Θα θέλαμε η Προεδρία σαφέστατα να διαβιβάσει στο Συμβούλιο την ανάγκη ύπαρξης σφαιρικής αντιμετώπισης και γενικής ισορροπίας του κειμένου. Διαφορετικά, θα είναι πολύ κρίμα για όλους και οι εισηγητέ που ήταν παρόντες σήμερα το απόγευμα και την Επίτροπο Μάλστρομ θα πρέπει να συνεχιστούν ακόμα περισσότερε συζητήσεις, κάτι που δεν είναι προ όφελο κανενό. Ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτής τη καταστάσεω. Δίνουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο, ο κ. Ματίας Ουλ, αν θέλετε έχετε το λόγο. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια καταρχήν για την πολύ επικοδομητική της προσέγγιση μέχρι τώρα που μας επέτρεψε να προχωρήσουμε πολύ σημαντικά. Μεγάλη πρόοδος από το Σεπτέμβρη όταν άρχισαν οι διαπραγματεύσεις ε, πάνω στο θέμα. Διευκρινήσαμε, βρήκαμε καταρχήν συμβιβαστικές λύσεις στα περισσότερα θέματα και όπως είπε και η κυρία Γκυλιόμ... αυτό έγινε σε ένα πολύ περίπλοκο θέμα ε, του πακέτου ασύλου συμφωνούμε και σε σχέση με το, την τελική φάση των διαπραγματεύσεων όπου χρειάζεται μια λεπτή και ισορροπημένη συμβιβαστική λύση. Εν ώψη των προβλημάτων πρέπει να βρούμε ένα πακέτο σχετικά με τα τελευταία εκρεμή θέματα. Δεν θα μιλήσω για τα εκρεμή θέματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί η κυρία Γκυγιόμ τα συνόψησε πολύ ωραία και λεπτομερέστατα. Από την πλευρά του Συμβουλίου, από εμά υπάρχει το δικαίωμα προσφυγής σε διαδικασίε συνόρων, μετέπειτα αίτησα, ε, ε, αίτηση και ανάκληση και για την Κομισιόν ήταν και είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί συμβιβαστική λύση που επαρκώς θα ε, προστατεύει θύματα βασανιστήριων και ασυνόδευτους ανηλίκους όπως αναφέρθηκε ήδη. Παράλληλα η Κομισιόν είναι έτοιμη να βοηθήσει για να βρεθούν κατάλληλες συμβαστικές λύσεις και σε όλα τα άλλα σημαντικά θέματα επίσης, ούτω ώστε στο τέλος να εξευρεθεί αυτή η ισορροπημένη συμβιβαστική λύση που θέλουμε. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το φάκελο, θα, ε, ο φάκελος συζητηθεί σε επίπεδο Α, εγώ περιορίζομαι σε αυτά που είπα. Ευχαριστώ. Από την Κυπριακή Προεδρία, ο κύριος Παπαγεωργίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, όπως είπε ήδη η εισηγήτρια, οι διαπραγματεύσεις για την οδηγία αυτή και συμφωνώ απόλυτα μαζί της, είναι οι πιο περίπλοκες, γιατί είναι το πιο σύνθετο θέμα για το άσυλο. Οι διαπραγματεύσεις πάντως προχώρησαν πολύ από το Σεπτέμβριο και τώρα μπήκαν στην τελική φάση, στο Προφανώς τα στοιχεία της τελικής συμβιβαστικής λύσης αρχίζουν σταδιακά και διαμορφώνονται. Ε, είμαστε, ε, έχουμε, ε, πιστεύουμε, όπως και η συγκήτρια, ότι είναι εφικτή η συμφωνία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι για το Συμβούλιο το τελικό κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες που θα είναι δίκαιες για τους ετούντες, αλλά που θα είναι και κοινέ ε, για τα κράτη-μέλη, λαμβάνοντας ε, παράλληλα υπόψη τα διαφορετικά δικαιικά συστήματα, αποφεύγοντας ε, άσκοπο διοικητικό φόρτο, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να εντοπίζουν καταχρηστικές πρακτικές. Έχουμε αμέσως και μια, συζήτηση, μια συνάντηση σχετικά με αυτό το θέμα. Εκείνο που θέλω να πω μόνο λοιπόν είναι ότι ε, η Προεδρία, το Συμβούλιο ε, είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί ε, ακατάπαυστα με την Επιτροπή για να βρεθεί μια λύση και είμαστε στο διάθεση της εισηγήτριας. Ευχαριστώ και την Κυπριακή Πρόεδρε για τη συμβολή τη, για τη συνεισφορά τη. Πολύ τριμερείς διάλογοι ε, λαμβάνουν χώρα. Έχουμε πέμπτο και έκτο γύρο που αναμένονται μετά τους τέσσερις που έχουν γίνει και επανερχόμαστε τώρα στην κυρία Κιγιόμ για τα τελικά συμπεράσματα της ε, σημερινής συζήτησης. Σε λίγο θα έχουμε τη συνάντηση της ε, ομάδας εργασίας που θα ασχοληθούμε με όλα αυτά τα θέματα. Δεν έχει νόημα να κάνω και άλλα σχόλια. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε αυτή την απογευματινή συνεδρίαση με μια ανακοίνωση εκ μέρους του συναδέλφου Κλοντ Μοράες, που διοργανώνει ε, μία ε, έκθεση και συζήτηση πάνελ για την ε, προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την, τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα αρχίσει στις 6.30, σε λίγα λεπτά δηλαδή, η συζήτηση πάνελ με διοργάνωση και υπό την του κ. Μωράες και ε, θα γίνει και μια δεξίωση για τα εγγένεια αυτής της έκθεσης ευκαιρία και της ετήσιας συνάντησης για την εξασφάλιση πρόσβασης στη δικαιοσύνη και καιρούς οικονομικής κρίσης. Για περαιτέρα λεπτομέρειε, ε, σα παραπέμπω στο γραφείο του κ. Κλοντ Μωράη που διοργανώνει αυτή την εκδήλωση και τη συζήτηση του πάνελ. Σε λίγο θα συνεδριάσει η διοργανική ομάδα επαφής για το άσυλο, φυσικά αυτό για τους ενδιαφερόμενους. Η τακτική συνεδρίαση τη Επιτροπής μας θα συνεχιστεί αύριο στι 9 σε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή νομικών υποθέσεων για κάποιες ψηφοφορίες που θα γίνουν για το πρόγραμμα δικαιοσύνης, άλλη όμως αίθουσα. Λύεται η συνεδρίαση.